welcome everybody to our LIBE meeting. I ask all the colleagues, members, assistants to take their seats, please. Σας παρακαλώ, καθίστε. Ας προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση μεταξύ, αρκετοί συνάδελφοι θα καταφτάσουν. So Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις. Προεδρεύω τη σας, διότι ο κανονικός πρόεδρος δεν μπορούσε να παρίσταται αλλά θα παρίσταται στην ε, αυριανή συνεδρίαση. το σημείο 16, η ψηφοφορία για τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα για την επιστροφή παρανόμως διμενών των υπηκών των τρίτων χωρών πρέπει να αναβληθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η τροποποιηθή σε μερισσία διάταξη. Δεν έχουμε διερμηνία στα κρατικά, και, δυστυχώς και στα αγολεδικά και σήμερα και αύριο. Να διαβάσω τις συστάσεις των συντονιστών που θα παρακαλούσα να εγκρίνεται διορισμός εισηγητών η κυρία Γκάμπρελ διορίστηκε εισηγήτρια για τα εξή θέματα εξαίρεση θεωρήσεων μεταξύ νήσων προδομώντας της Ευρωπαϊκής Ανώσης Μικρονησία του Βαλού και νήσων Μάρσαλ για παραμονή μικρής διαρκείας διορίστηκε η συγγήτρια για μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό που παραθέτει τις τρίτες χώρες των οποίων οι πίκοοι θα πρέπει να έχουν θεωρήσεις όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα και εκεί είναι στις χώρες οι πίκοοι των οποίων εξαιρούνται από την απέτηση αυτή. Ο κ. Δίας Δεμέρεα διορίστηκε ως εισηγητής για μια πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό που παραθέτει τι χώρε υπήκοοι των οποίων θα πρέπει να έχουν θεωρήσει όταν διέρχονται εξωτερικά σύνορα και τι χώρε εκείνε ε, των οποίων υπήκοοι εξαιρούνται από αυτέ τι απαιτήσει, αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολή, αντί αυτή περίπτωση. Η κυρία Φαϊγιόν διορίστηκε σαν εισηγήτρια για μια πρόταση κανονισμού που παραθέτει τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι θα πρέπει να έχουν θεωρήσει όταν διέρχονται εξωτερικά σύνορα και τις χώρες εκείνες που εξαιρούνται από αυτή την απέτηση. Το κοσυφοπέδησε την περίπτωση. Ο κύριος Νίντερ είναι συγγητής για την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το άσυλο και την αστολή του κανονισμού 439 του 2016. Η κυρία Κανίτσι είναι η συγγήτρια για γνωμοδότηση για την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την καταπολέμηση της απάτης. Η Επιτροπή Κόντι είναι η καθήλυνα αρμόδια. Αυτά, αυτές λοιπόν ήταν οι συστάσεις των συντονιστών για τις διάφορες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Εγκρίνεται τις συστάσεις αυτές. Θεωρώ ότι συμφωνείτε. Έχουμε έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 25ης Απριλίου και 1ης Οκτωβρίου του 2016 και 1ης Οκτωβρίου του 2015. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά θεωρούνται συγκεκριμένα και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεώς μας. Έχουμε λοιπόν συζήτηση επί του σχεδίου εκθέσεω και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το πρωτόκολλο να εξαλειφθεί το παράνομο εμπόριο των προϊόντων καπνού στα πλαίσια του ΠΟΕ για, τον, για τη Σύμβαση για τον Έλεγχο των Προϊόντων Καπνού όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που εμπίπτουν στο κατηγορία 5 του τρίτου τμήματος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σχετικά με αυτά λοιπόν, μετά τις συστάσεις της εισηγήτριας, της κυρίας Άντερσον, που θα καταφθάσει αργότερα, ήρθε σε επαφή με τη γραμματεία, μας ειδοποίησε, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση εν τη απουσία της, θα καταφθάσει αργότερα. Λοιπόν, πρότεινε και οι συντονιστές συμφώνησαν να ανταλλάξουμε απόψεις με τους εκπροσώπους της ε, Όλαφ και της DG Sante. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Ρόμπλινγκ τη Όλαφ και στον κύριο Μπορκόφσκι μετά τη DG Σάντε και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση ο κύριος Ρόμπλινγκ λοιπόν έχει το λόγο ορίστε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα λέει και ο Ζρόμπλινγκ, ακόμα και αν δεν είναι εδώ η συγγήτρια, ξεκινώ συγχαίροντά την. Η κυρία Άντερσεν έκανε έξοχη δουλειά. Και σύντομα μάλιστα στον φάτο το σχέδιο συστάσεως τη. Είναι δίκαιο να πούμε ότι το παράνομο εμπόριο καπνού μας προβληματίζει πολλού. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν δισεκατομμύρια από έσοδα κάθε χρόνο το λαθρεμπόριο υπονομεύει και τις πολιτικές τιμολόγησης ε, που τίθενται προς όφελος της ε, υγείας, της δημόσιας Τα τσιγάρα γίνονται πιο προσβάσιμα και για τους νέους μέσω του παρανόμου εμπορίου. Και το λαθρεμπόριο είναι μεγάλη πηγή εισοδημάτων για το οργανωμένο έγκλημα. Τι κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι περίπλοκο φαινόμενο. Και δεν υπάρχει μία λύση που από μόνη σας σταματήσει το φαινόμενο. Τι πρέπει να κάνουμε. Να αναθερούμε συνεχώς την εργαλειοθήκη μας και να δούμε τα εργαλεία μας είναι τα καλύτερα. Μπορούμε στο βαθμό του δυνατού να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο σιγαρέτων. Έχοντας αυτό υπόψη, πριν από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα έγγραφο στρατηγικής. Καθορίζει ανάλυση και διεξόδους για την αύξηση τη καταπολεμής του εθρομπορίου σιγαρέτων. Είμαστε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, στενή συνεργασία, εφαρμόζοντα καθημερινά αυτή τη στρατηγική. Σε αυτό συμπεριλαμβάνουμε επιχειρησιακά μέτρα, έρευνε, νομοθεσία, όπως αυτή που έχουμε μπροστά μα, και ένα ευρύ φάσμα πολιτικών. Εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, εδώ και δύο χρόνια, έχουμε την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Συμπεριλαμβάνουν τι διατάξει όσον αφορά την ιχνηλάτηση των προϊόντων. Εμείς στο Όλαφ, στην Όλαφ, ανησυχούμε τα μάλα για το λαθρεμπόριο σιγαρέτων από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά αυτά τα σιγαρέτα. Σχετικά με αυτό, το νέο πρωτόκολλο που συζητούμε σήμερα εδώ, είναι μια ρηξικέλευτη πρωτοβουλία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πολυμερή πρωτοβουλία. Καλύπτει σφαιρικά το πρόβλημα του λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με υπερηφάνεια θα λέει που ηγείται στη διαπραγμάτευσή του μέσω αυτού και με τις προσπάθειες αυτές την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ανάλυση στο Συμβούλιο και ελπίζουμε τελικά και με τη συνένεση του Κοινοβουλίου μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε αποφασιστικοί για να εγκρίνουμε, να, να κυρώσουμε αυτό το μέσο. Καλωσορίζουμε τη στήριξη των κρατών μελών στο Συμβούλιο για το έγγραφο και ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα προχωρήσει στην όλη διαδικασία κύρωση Για λόγους νομικούς πρέπει η σύσταση να χωριστεί σε δύο ξεχωριστά έγγραφα. Ξεχωριστά αλληλένδετα βέβαια όμως. Βλέπουμε τα χαρά ότι η Επιτροπή Ίντε ήδη ομοφόνος από ό,τι καταλαβαίνω στήριξε το άλλο έγγραφο σας. Τώρα το δεύτερο το έχουμε σήμερα μπροστά μας και θέλω να στηρίξουμε το σχέδιο συστάσεως που υπέβαλε η συγγήτρια και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούμπλινγκ. Ο οποίο Μπολκόφσκι. Thank you, ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ε, απόλυτα με την παρουσίαση του εκπροσώπου της ΟΛΑΒ, γιατί και η Γενική Διεύθυνση της Υγεία ε, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό, το πρωτόκολλο, και εμείς με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού έχουμε το άρθρο 15, που θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τον αντοπισμό και την ανείχνευση. Είναι μία από τις βασικές διατάξεις και του πρωτοκόλου και το εφαρμοστικό έργο που ασκούμε θα ε, οδηγήσει μέχρι την 20 Μαΐου του 2019 την εγκαθίδρυση του συστήματος και μάλιστα ε, τη διορία τη βάζει το πρωτόκολλο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί αφορά την έμπρακτη εφαρμογή του πρωτοκόλλου και μάλιστα παγκοσμίω. Γι' αυτό και εμείς θα πρωτοστατήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και ευχαριστώ θερμά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δική του πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπορκόφσκι. Πάνω στην ώρα ήρθατε κύριε Άντερσον. Μόλις ε, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της ΟΛΑΦ, τον κύριο Ρούμπλινγκ, και τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΤΕ, τον κύριο Μπορκόφσκι, μας έκαναν πολύ σύντομες παρεμβάσεις για το θέμα αυτό. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Άντερσον, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Μάλιστα και σας ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Χθε το απόγευμα σε έξι έφυγα από το σπίτι μου, ελπίζοντας να έρθω εγκαίρωση. Και εξαιτία των δύο καθυστερήσεων που είχα συμπτήσει, κατάφερα και έφτασα καθυστερημένα. Παρά τι προσπάθειε που έκανα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το τσιγάρο σκοτώνει κάθε χρόνο 6 εκατομμύρια ανθρώπου. Γι' αυτό και είναι σημαντική η ακρόαση που οργανώσαμε. Και μάλιστα ε, είναι τοξική αυτή η ουσία. Και το γνωρίζουμε ήδη ε, εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης, ε, έχουμε το πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το λαθρεμπόριο των προϊόντων καπνού. Αυτό συζητούμε σήμερα. Και το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άντε και τη ΟΛΑΦ για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και των συναφών άρθρων είναι χαρακτηριστικό. Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να ε, διασφαλιστεί η προστασία όλης της αλυσίδας ανεφοδιασμού προϊόντων νόμιμων προϊόντων καπνού και μάλιστα θα πρέπει να καταβάλλονται και οι τελωνιακοί δασμοί και να πληρούνται όλε οι καθ' ε, καθόλου του κρίκου τη αλυσίδα του ανεφοδιασμού καπνού. Το άρθρο αυτό του πρωτοκόλου υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να θεσπίσουν ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού και ανείχνευση ε, μέσα σε μια πενταετία από τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλου. Και πρόκειται για μια παγκόσμια λύση ε, διεθνούς εμβέλειες γιατί το πρόγραμμα είναι διεθνές και ε, τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εγκρίνουν το πρωτόκολλο. Βέβαια, έχουμε ανησυχίες και προβληματισμό για τη σχέση με την βιομηχανία, την καπνοβιομηχανία, ε, που δημιουργεί κάποια προσκόμματα στην ευόδοση της έγκρισης του πρωτοκόλλου. Παρά είναι φιλική σχέση ευρωπαϊκή Ένωσης και καπνοβιομηχανία. Βλέπουμε την καπνοβιομηχανία ε, σαν ε, φίλο, συμβαλόμενο μέρος, ενώ ε, το 2008 είχαμε τέσσερις καπνοβιομηχανίες που καταδικάστηκαν γιατί συμμετείχαν κατά κάποιο τρόπο στο λαθρεμπόριο καπνού, γιατί δεν, είχε, δεν ήταν συσκευασμένα τα προϊόντα, δεν είχαν ε, ούτε σφραγίδα και ε, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Έγιναν έρευνες από την Όλαφ και μάλιστα η GTI Tobacco International κα, κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο τσιγάρων στη Μέση Ανατολή και είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας σήμερα, παρόλο που δυστυχώς έχασα την σύντομη παρουσίαση που κάνατε στην αρχή. Ελπίζω να με ενημερώσει ε, οι συνεργάτε μου, οι μου για αυτά που είπατε και πώ ενημερώσατε του συναδέλφου για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Γιατί ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και ιδιαίτερα το λαθρεμπόριο τσιγαρέτων που εξάγονται σε περιοχέ που δεν έχουν σαφώς ρυθμισμένη αγορά. Και ε, επανέρχονται μέσω αυτών των ε, δικαιοδοσιών πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα μερικέ ε, παράνομα τσιγάρα είναι γνωστό, γνωστών μαρκών που κάπου ε, μέσα στο σύστημα διαμετακόμισης ε, χάνονται ως διαμαγείας. Επίσης αυτά τα blue white, τα ε, τσιγάρα χωρίς μάρκα είναι νέα προϊόντα της αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να, να μας πείτε τι έγιναν μετά τα πορίσματα και του διαμεσολαβήτη. Τι έγινε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εφαρμοστεί το άρθρο 5,3 του τη ύφεση για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού. Και τι θα κάνει η Γενική Διεύθυνση Σάντη για όλα αυτά, γιατί η Philip ε, ε, Morris International έχει συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του λαθρεμπόριου καρπού και παρόλα αυτά θα πρέπει, δεν πληρεί τις υποχρεώσεις για τον εντοπισμό και ανείχνευση των παρανόμων τσιγάρων. Είναι σαν να βάζουμε το λίγο να φυλάει τα πρόβατα δίνοντας τέτοιες εξουσίες στη Φίλιπ Μόρις. Και μάλιστα πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχίε για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ε, ηγετικό στέλεχος του Φίλιπ Μόρις ότι έχουμε κοινούς στόχους για την, με τη σύμβαση πλαίσιο για να πατάξουμε το παράνομο εμπόριο, το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Κάτι που απάδει από την ε, αλήθεια και την πραγματικότητα. Γιατί ε, φαίνεται ότι οι καπνοβιομηχανίες ε, εμποδίζουν παγκοσμίω πολλές χώρες να, να προσυπογράψουν το πρωτόκολλο. Και σίγουρα αυτή η δήλωση είναι αναλυθής. Και μάλιστα το 2004 είχαμε κάποιες αγωγές που καταδικάζουν και καταγγέλουν την ε, συμμετοχή της ε, καπναβιομηχανίας στο παράνομο εμπόριο. Και μάλιστα η Φίλιπ Μόρις μέχρι στιγμής ε, εξαιτία αυτού έχει καταβάλει 1,1 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα δεν το έκανε καθόλου από αγαθοεργία ή από φιλανθρωπικό σκοπό. Ήταν ένας συμβιβασμός νόμιμος. Και παρόλα αυτά η σύμβαση πλαίσιο και τα πρωτόκολλα τα λένε καθαρά ότι η καπνοβιομηχανία είναι τμήμα του προβλήματος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα της λύσης. Και πρόκειται αναφεσβείται, για ένα πεδίο μάχη. Στη μία πλευρά βρίσκεται η καπνοβιομηχανία και η σύμβαση του ΠΟΗ από την άλλη πλευρά. Έχουμε τα άρθρα 8,12 που δεν αναφέρονται ή ε, το άρθρο 5 παράγραφο 3 που προβλέπουν το σαφή διαχωρισμό που πρέπει να γίνει μεταξύ της καπνοβιομηχανίας αφενός και όλων των υπόλοιπων αφετέρου. Και ιδιαίτερα αναφέρεται η σχέση που θα πρέπει να υπάρχει για την ανάπτυξη πολιτικών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται η καπνοβιομηχανία. Πάνω από 100 συμβαλόμενα μέρη ανά τον κόσμο έχουν ε, προσυπογράψει τέτοιες ε, προαιρετικές συμφωνίες με την καπνοβιομηχανία που αναφυσβήτητα κατά τη γνώμη μου ε, διακυβεύουν τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλου της Παγκοσμίας Οργάνωσης Υγείας. Εγώ είμαι υπέρμαχος του πρωτοκόλου και έχω σοβαρές ανησυχίε για το σύστημα ε, που ε, έχει εφαρμόσει με τη Φίλιπ Μόρις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το σύστημα αυτό δεν ε, εξυπηρετεί καθόλου, δεν καθόλου το σκοπό της ενίχνευσης και εντοπισμού των προϊόντων καπνού. Και μάλιστα υπάρχει ένα black box που πρόσφερε η καπνοβιομηχανία που δεν ξέρουμε καν το περιεχόμενό, μου, το περιεχόμενό του και σίγουρα ο έλεγχος ε, που θα εξασφαλίσει η καπνοβιομηχανία δεν είναι επαρκής. Θέλει να μας αυτοπαρουσιαστεί ως ε, υπεύθυνο ε, μέρος απέναντι στα κυβερνητικά όργανα, αλλά νομίζω ότι δεδομένες και της έρευνας της Όλαφ έχουμε σαφείς αποδείξει και τεκμήρια για το ότι δεν είναι σοβαρή εταίρη. Και μάλιστα και μετά την οδηγία για το περίοδο καπνού έχουμε πολλέ αμφιβολίε ε, για το ρόλο που έπαιξε μέχρι στιγμή η καπνοβιομηχανία. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα για το θέμα αυτό, αλλά με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η άποψη και των συναδέλφων και κυρίω οι πληροφορίε τη ΟΛΑΦ και οι περαιτέρω διευκρινήσει για την πορεία των ερευνών που έχει κάνει σε σχέση με τις καταγγελίες και κατηγορίες κατά της καπνοβιομηχανίας. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούει και προσέχει τα πορίσματα του διαμεσολαβητή που λέει ότι για να προασπιστεί η δημόσια υγεία δεν θα πρέπει να ευθύνεται μόνο μία μόνο Γενική Διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Είναι συλλογική ευθύνη ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Επίση, ε, θα ε, εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτόκολλο. Θα το κυρώσει. Τι γίνεται με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καπνοβιομηχανιών που θα λήξει τον Ιούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπερψηφίσει πρόταση, ψήφισμα, για τη μη ανανέωση της συμφωνία αυτή με την καπνοβιομηχανία. Θα εισακουστεί η επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διακοπεί επιτέλου αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Ο λόγο στον κύριο Σόγκρο, σκιώδη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Το παράνομο εμπόριο καπνού δεν δημιουργεί μόνο απώλειες στα έσοδα των κρατών μελών, αλλά παραβιάζει και τις πολιτικές δημόσιας υγείας των κρατών μελών και τις πολιτικές που αφορούν την διανομή των καπνικών προϊόντων. Ε, πρέπει να ε, αποτραπεί η δυνατότητα παράκαμψης των πολιτικών που έχουν θεσπιστεί ο έλεγχος λοιπόν της ε, αλυσίδας εφοδιασμού είναι σημαντικός όχι μόνο για τον έλεγχο των ε, προϊόντων αυτών καθ' αυτών, αλλά και για την μείωση της χρήσης προϊόντων καπνού. Αποδεικνύεται ε, από τα στοιχεία ότι τα παράνομα τσιγάρα πολλές φορές καταλήγουν και μέσω διαφόρων διάβλων στην αγορά. Και υπάρχει μεγάλο περιθώριο κερδοφορίας στα παράνομα τσιγάρα. Ε, υπάρχει, δυνατότητα μεγάλης κάλυψης του κόστους παραγωγής των προϊόντων μέσω της παράνομης διάθεσης τους στην αγορά. Και όπως ε, δείχνει και μια περίπτωση του Όλαφ, που διερεύνησε Όλαφ το 1998, ε, παραγωγός κατάφερε ε, τσιγάρων κατάφερε να υπερκεράσει το, το κόστος ε, που είχε επομιστεί για την παραγωγή μιας ποσότητας τσιγάρων δεν μπορούσε όμως να αποδείξει από πού, είχε, που, πού είχαν προέλθει οι πόροι για την παραγωγή των τσιγάρων αυτών. Όπως ε, αναγνωρίζεται και στην νέα στρατηγική για την ασφάλεια που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν το 2015 αναγνωρίζεται το πρόβλημα λόγω και της ε, γκρίζας αγοράς που κυριαρχεί στον τομέα αυτών, όλα, όλα αυτά τα στοιχεία ε, αποτελούν απλώς εκτιμήσεις και σε, στην καλύτερη περίπτωση, ε, από ό,τι φαίνεται, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού διακινούμενου όγκου. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και συντονισμένη παγκόσμια αντίδραση και ρύθμιση του παράνομου εμπορίου καπνού. Καλό νέο είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό επίπεδο παράνομου εμπορίου δεν ε, συνδέεται με την ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και ότι τα κράτη-μέλη μπορούν, ε, έχουν ενισχυμένα εργαλεία στα χέρια τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, στην μελέτη σκοπιμότητας της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε τον περσινό Μάιο, ε, αποδεικνύεται ότι υπάρχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και εχνηλάτησης των προϊόντων καπνού και ότι σε όποια, όποια επιλογή και αν ε, γίνει ε, τα πλεονεκτήματα θα υπερτερούν των μειονεκτημάτων. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης. Το άρθρο 15 της αναθεωρημένης οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα ήδη προβλέπει τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος με την δημιουργία ε, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που θα επιτρέπει αυτή την παρακολούθηση και ανείχνευση. Και το άρθρο 8 ε, του πρωτοκόλου συνάδει ακριβώς με αυτό το σύστημα παρακολούθησης και ανείχνευσης. Ωστόσο, ε, καθώς σημαντικό μέρος της παραγωγής ε, παράνομων τσιγάρων προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται και διεθνή συνεργασία. Το πρωτόκολλο είναι η καλύτερη απάντηση πολιτικής στο διασυνοριακό πρόβλημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ακριβώς διότι προβλέπει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης της ανείχνευσης και της παρακολούθησης του ξεπλήματος ε, χρήματος ε, και της ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να βοηθήσει ε, στην εξασφάλιση της ακαιρεότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά θα πρέπει να βασίζεται και σε μέτρα δίωξης, διερεύνησης και διεθνούς συνεργασίας στο δικαστικό τομέα. Η ταχεία κύρωση του πρωτοκόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη ακριβώς διότι μεταξύ άλλων θα δώσει στα 28 κράτη-μέλη και σε άλλες χώρες ε, ε, ε, τη δυνατότητα να έχουν ένα τέτοιο εργαλείο νομικά δεσμευτικό στη διάθεσή τους. Η κυρία Γκόμες, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, ιδιαίτερος την εισηγήτριά μας αλλά και τον κύριο Σόγκαρ για την συμβολή και τη βοήθειά του στην εισηγήτρια. Θα ήθελα να προσθέσω λοιπόν ότι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο που δεν έχει εξεταστεί ε, επαρκώς λόγω και του επίγοντος χαρακτήρα των δραστηριοτήτων μας είναι ότι υπάρχει σημαντική σύνδεση μεταξύ των δικτύων οργανωμένου ε, εγκλήματος όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην ε, ευρύτερη γειτονία μας και ιδίως στην ε, Βόρεια Αφρική που συνδέεται με τα δίκτυα αυτά λοιπόν συνδέονται και δραστηριοποιούνται στην διακίνηση παράνομων τσιγάρων αλλά και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων και βεβαίως την τρομοκρατία. Κάτι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το παραβλέπουμε. Αντιθέτως, ε, επιτείνει την ανάγκη να αναλυφθεί δράση και ε, ε, συμφωνώ και εγώ με την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός με την DG εσωτερικών υποθέσεων και τον ε, Ευρωπαίο Συντονιστή για την καταπολέμηση της Θερμοκρατίας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευθυνθεί και να, αναλάβει εκείνα τα, λάβει εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την ε, διακοπή της ροής παράνομων ε, προϊόντων ε, ένα θέμα στο οποίο η καπνοβιομηχανία πράγματι παίζει σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω και εγώ την εισηγήτρια. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει αναφυσβήτητα προκαιρού. Στην Ευρώπη έχουμε ιστορικών εκπροσώπων, υψηλά σταμένων εκπροσώπων των 100 μελών που έπρεπε να παραιτηθούν λόγω κατηγοριών για παράνομες δραστηριότητε. Ξέρουμε ότι το παράνομο εμπόριο των ε, καπνικών προϊόντων ε, είναι κάτι πραγματικό, συμβαίνει καθημερινά σε όλη την Ευρώπη. Οπότε το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί το ταχύτερο δυνατόν, σε πλήρη διαφάνεια και εμείς σαν ομάδα το υποστηρίζουμε πλήρως. Επίσης, θέλω να πω ότι η καπνοβιομηχανία ίδια έχει ευθύνε. Πρέπει να αναλάβει τη δέουσα δράση, ούτω ώστε άπαξ απαντός να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο των καπνικών προϊόντων. Όλα τα μέρη λοιπόν, τα συμβαλόμενα του πρωτοκόλου, θα πρέπει να κινηθούν διαφανώς σε πλαίσια διευρυμένης συνεργασίας με την καπνοβιομηχανία. Και όταν θέλουμε να προβούμε στην ανείχνευση της προελεύσεως των προϊόντων, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου την εισηγήτρια. Έκανε έξοχη δουλειά. Και ας ελπίσουμε ότι στην Ευρώπη πραγματικά θα υπερασπιστούμε αυτή τη θέση. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ κυρία Βίκστρομ. Ο κύριος Ρόμπλινγκ ξανά έχει το λόγο, ο εκπρόσωπος της ε, Όλαφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχωρήστε με καταρχάς αν επαναλάβω κάτι. Δεν ήταν παρούσα η συγγήτρια πριν από μισή ώρα και ζητώ συγγνώμη που ξεκίνησα την παρουσίαση της εκθέσεως, των σχολιασμών της εκθέσεως τη. Ζητώ συγγνώμη και επαναλαμβάνω την πρώτη μου φράση. Θέλω να τη συγχαρώ, σα σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε τάχιστα ε, για αυτή την έκθεση και ότι είναι πολύ καλή η έκθεση. Τόσο αφορά τα θέματα που ετέθησαν, να πω το εξή. Όσον αφορά την ανείχνευση, η χνηλάτιση, στα πλαίσια της οδηγίας των προϊόντων καπνού, όλα αυτά θα τα απαντήσει καλύτερα ο άνωθεν συνάδελφος ο Τουσιππίν της Γενικής Διευθύνσεως Υγείας, διότι αυτή η υπηρεσία ασχολείται με το θέμα αυτό της ε, ηχνηλάτης προελεύσεως των προϊόντων και ίσως μετά από μένα ο συνάδελφος να μιλήσει διότι ίσως ε, θα μπορέσει να προσθέσει κάτι στα σχόλιά μου. Τώρα, απαντώντας σε αυτά που ετέθησαν, χαίρομαι διότι περισσότεροι στην αίθουσα συμφωνούν ότι είναι σημαντικό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Τρίτον, το πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα χρειάζεται μια σφαιρική απάντηση και το πρωτόκολλο είναι η καλύτερη απάντηση. Πρέπει να χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παρελθόν ηγήθηκε στις διαπραγματεύσεις για αυτό το μέσο. Και υπάρχει και συνένεση που διαμορφώνεται και προσβλέπουμε και στην κύρωση του εν λόγω μέσου. Διάφοροι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν την αλλαγή της φύσεως του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε με αυτό. Ένα έγγραφο στρατηγικής, συνετάχθη προτριετίας. Εκεί τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων σήμερα έχει διαφορετική μορφή από ό,τι πριν από 10-15 χρόνια. Κατά το παρελθόν η αγορά κυριαρχεί το από από πραγματικά ε, προϊόντα και από παραπημένα προϊόντα. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Αν δούμε τις κατασχέσεις των κρατών μελών, στην καθημερινή μάχη που δίνουν τα κράτη-μέλη, βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα κατασχόμενα σιγαρέτα είναι από τις ανώνυμες εταιρείες. Έχουν ένα όνομα, αλλά τέλος πάντων τα κατάσχονται καθημερινά αυτά, τα ανώνυμα το ΣΥΠΗΝ. Πέρσι, Φερρυπίν, η Όλαφ έσπασε ρεκόρ του όγκου των τσιγαρέτων που κατασχέθηκαν με τη βοήθεια της Όλαφ στα κρατη Υποστηρίξαμε περίπου την κατάσχεση 600 εκατομμυρίων τσιγαρέτων. Κάθε ένα τσιγάρο αυτό ήταν τα cheap whites. Στατιστικά, αν έχουμε ένα πακέτο σιγαρέτων με 20 σιγαρέτα, εμείς συμβάλαμε σαν όλα στατιστικά να κατασκευθούν 3 με 4 σιγαρέτα παράνομα από αυτό το πακέτο. Συμφωνούμε. Είναι σημαντική η αύξηση της προσπάθειας κατά πολεμήσεως του φαινομένου. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε αργότερα αυτό το έτος να υποβάλει έκθεση. Η έκθεση αφορά την εφαρμογή του εγγράφου του 2013. Νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο έγγραφο θα τονίζεται ιδιαίτερα το φαινόμενο των Chip whites, αυτό των ανωνύμων σιγαρέτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ παρανόμου εμπορίου καπνικών προϊόντων, προϊόντων που έρχονται απ' έξω από το εξωτερικό, μαζί με, και τη σχέση που έχει αυτό με το ε, οργανωμένο έγκλημα. Καθημερινά και εβδομαδία συνεργαζόμαστε με την DG Home, ανταλλάσσουμε απόψει. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι στην καταπολέμηση του φαινομένου για να είμαστε αποτελεσματικοί. Συζητούμε με τη Frontex, την Europol και με άλλου φορεί και με τα κράτη-μέλη βέβαια. Υπάρχει συνεργασία. Για το θέμα Philip Morris, θα ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου υπέβαλε ένα έγγραφο τεχνικής αξιολογήσεως. Συζητήθηκε εκτενώς στο Κοινοβούλιο και στις 9 Μαρτίου το Κοινοβούλιο ψήφισε, πέρασε μάλλον ένα ψήφισμα. Εμείς εξετάζουμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα. Για το άρθρο 5,3 παραπέμπω στη γραπτή απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απεστάλει στο διαμεσολαβητή και δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτή την απάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις κύριε Ρούμπλινγκ. Ο κύριος Μπορκόφσκι. σε ό,τι αφορά το εφαρμοστικό έργο, σε ό,τι αφορά το σύστημα παρακολούθηση και ανείχνευση στην Ευρώπη, αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι συνεχίζεται αυτό το έργο εφαρμογή. Δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα πώς, ε, το πώ θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω στο μέλλον το σύστημα αυτό παρακολούθηση και ανείχνευση. Πάντω, ε, εμεί ε, θεωρούμε ότι το πρωτόκολλο θα κυρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ. Με αυτό το σενάριο συνεχίζουμε τις δικές μας εργασίες και αναπτύσσουμε αυτό το σύστημα παρακολούθησης και ανείχνευσης που θα ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Υγείας. Για παράδειγμα, το άρθρο 8.2, 8.12. Βέβαια δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με όλα τα άρθρα και τις παραγράφους του πρωτοκόλλου. Το άρθρο 8.2 απαιτεί έλεγχο του συστήματος από τα συμβαλόμενα μέρη εμπροκειμένου προκειμένου το δικό μας σύστημα θα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 8.12 του πρωτοκόλλου υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να μην εχωρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στην καπνοβιομηχανία. Είχαμε επαφές με την καπνοβιομηχανία προκειμένου να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα παρακολούθηση και ανείχνευση. Η ανάμειξη όμω τη καπροβιομηχανία στην ανάπτυξη αυτού του συστήματο ε, θα περιορίζεται στο απολύτω απαραίτητο, όπω προβλέπει και το πρωτόκολλο, να μην εκχωρηθούν οι δικέ μα υποχρεώσει στην καπροβιομηχανία. Μόνο που είναι απολύτω απαραίτητο και στα πλαίσια τη εφαρμογή του άρθρου θα έχουμε κάποιε ανάληψη υποχρεώσεων και από την καπνοβιομηχανία. Και σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει από τρίτο μέρος. Ε, χρειάζεται μία επαφή αλλά το σύστημα παρακολούθησης και ανείχνευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πλήρως ανεξάρτητο και θα παρακολουθείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο και όχι ε, από την καπνοβιομηχανία, ούτε θα ανατεθεί στα χέρια της καπνοβιομηχανίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Άντερσον, χρόνο φίδο παρακαλώ. Ε, μάλιστα, χαιρετίζω τα σχόλιά σας και ιδιαίτερος ε, το τελευταίο σχόλιο του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης ε, Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που εξάγω εγώ από το σχόλιο σας είναι ότι δεν χωρεί παράταση της συμφωνίας με τη Φιλίπ Μόρις, γιατί το σύστημα παρακολούθησης και ανείγνευσης ε, θα τηρεί πλήρως ε, και θα συνάδει με τις διατάξεις του πρωτοκόλου. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί το άρθρο 8 του πρωτοκόλου του ΠΟΗ ε, λέει ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων ε, και ιδιαίτερα στο 2 και 3 αναφέρεται ότι κάθε σεβαλόμενο μέρο ε, με βάση το άρθρο αυτό θα εγκαθιδρύσει ένα σύστημα παρακολούθηση και ανείχνευση που θα ελέγχει το ίδιο το συμβαλόμενο μέρο για όλα τα προϊόντα καπνού που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην επικράτειά του. Οπότε δεν νοείται εδώ να αναλάβει η καπνοβιομηχανία το σύστημα παρακολούθηση και ανείχνευση όπω συνέβαινε στο παρελθόν και κάτι και μάλιστα αυτό μα δημιούργησε τεράστιε ανησυχίε και προβληματισμό. Χαίρομαι για τι δηλώσει του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει τα ενία αποκλειστικά αυτού του συστήματο παρακολούθηση και ανείχνευση και επίση χαίρομαι που και ο ΛΑΒ προωθεί την κύρωση του πρωτοκόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αναφίβολο ότι χρειάζεται η επικύρωση αυτού του πρωτοκόλου και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Και δεδομένη τη συνένεση που έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε, από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, έχουμε μια ισχυρή εντολή να προωθήσουμε αυτό το θέμα και να επιτύχουμε την κύρωση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ και τους και οδησηγητές για τα σχόλιά σας και ευελπιστώ ότι θα προωθήσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Άντερσον. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στις 24 Μαΐου λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και με βάση το άρθρο 99.1 ε, του εσωτερικού κανονισμού, οι τροπολογίες ε, ε νο, ε, γίνονται δεκτές μόνο αν θέλουν να μόνο στο μέτρο που δεν αναθεωρούν τις συστάσεις του εισηγητού. Η έγκριση της έκθεσης θα γίνει στις 30 Μαΐου. επαναλαμβάνει 24 Μαΐου λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας, Ρούμπλινγκ και Μπορκόφσκι. Ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Άντερσον και περνάμε αμέσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας της Επιτροπής ΚΟΣΗ. Πρόεδρος της είναι ο κύριος Έιζερμαν. Όπως γνωρίζετε, η μόνιμη αυτή επιτροπή, η ΚΟΖΗ, εμ, συστήθηκε με βάση το άρθρο 71 της συνθήκης προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και να προωθεί συντονισμός και ανάληψη δράσης από τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και πολύ σημαντική Περιμένουμε λοιπόν την παρουσίαση του Προέδρου της Επιτροπής Κόζη. Καλώς ήρθατε κύριε Έζερμαν και θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τις δραστηριότητες της μόνιμης Επιτροπής σας και για τα μελλοντικά της σχέδια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να, για να έρθω να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητε της ΚΟΖΗ, της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση για τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της ΚΟΖΗ που έχετε λάβει και που καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2014 έως Δεκεμβρίου 2015. Προτού το κάνω αυτό όμως, θα άξιζε τον κόπο να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα σχετικά με την ε, μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Επιτροπή αυτή, η ΚΟΖΗ, με σκοπό την ε, πολυδιάστατη ε, μεθοδολογική προσέγγιση για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για τον ε, ε, κύκλο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται από τέσσερα βήματα. Πρώτο βήμα είναι η ευρωπαϊκή αξιολόγηση απειλής για, σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Σόκτα βασίζεται σε στοιχεία της Europol, ανάλυση των ε, κινδύνων και απειλών και συστήνει ε, ορισμένες ε, κατευθύνσεις γραμμές για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεύτερο βήμα στη συνέχεια είναι τα πολυετή στρατηγικά σχέδια που αναπτύσσει η ΚΟΖΗ, η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και οργανισμοί όπως η Frontex, η Europol και υπάρχει πολιτές στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένες προτεραιότητες και αυτά τα σχέδια ε, εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Τρίτο βήμα είναι τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης που ε, κατανέμονται αναέτος και αναπροτεραιότητα, συντάσσονται από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, σε αυτά τα σχέδια δράσης και εγκρίνονται από την ΚΟΖΗ. Και η Impact, το η ευρωπαϊκή ε, πολυδιάστατη πολυτομεακή ε, ε, πλατφόρμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έχει την έδρα της και γίνεται ο συντονισμός αυτού με ευθύνη της Europol. Η Europol λοιπόν υποστηρίζει αυτήν την πλατφόρμα και η COSI παρακολουθεί τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων. Και τέταρτο βήμα είναι η αξιολόγηση που ε, θα γίνει ε, τώρα το 2016 όπως αναφέρεται στην έκθεση και που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των κρατών μελών προκειμένου να αντιληφθούν διδάγματα για την, ε, τον επόμενο κύκλο πολιτικής. Πέρα από την έκθεση που σας αποστήλαμε θα ήθελα να σας, να σας ενημερώσω για τα θέματα που συζητήθηκαν επί Ολλανδικής Προεδρίας και που έθεσε και ο Υπουργός, ε, ο Ολλανδός Υπουργός κατά την έναρξη της Ολλανδικής Προεδρίας σε εσά. Η ενίσχυση της συνεργασίας, της επιχειρησικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων της ΚΟΖΗ και οι ε, αποτρόπες επιθέσεις στις Βρυξέλλες 22 Μαρτίου βεβαίως ενίσχυσαν για άλλη μια φορά την ε, την ανάγκη να ε, ενισχυθεί η συνεργασία μας και η ανταλλαγή πληροφοριών. Οι βασικές μας ε, ε, αξίες που επλήγησαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις πέρσι και φέτος είναι αυτές που βρέθηκαν στο επίκεντρο. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην ε, υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, της ιδιωτικότητας αφενός και αφετέρου της δίωξης και της καταδίκης ε, τρομοκρατών από την άλλη πλευρά. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών είναι απόλυτη προτεραιότητα ε, για την ε, Προεδρία από την έναρξη της υπάρχει ανάγκη να μετακινηθούμε σε μια ενιαία αντίληψη και μια βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και χρήση συστημάτων. Γι' αυτό το λόγο ε, χρειάζεται να ε, καταρτήσουμε έναν οδικό χάρτη που θα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αφορά την επιβολή του νόμου, τον έλεγχο των συνόρων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι διαπραγματεύσει βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να, σας να παρουσιάσουμε αυτόν τον οδικό χάρτη στο Συμβούλιο Τζάι στις 9 και 10 Ιουνίου. Αυτή... Αυτός ο οδικός χάρτης επίσης συνδέεται και με την ανακοίνωση της Κομισιόν για την ε, ε, για τα έξυπνα συστήματα και τον έλεγχο των συνόρων που παρουσιάστηκε 26 Απριλίου. Βλέπετε στην έκθεση ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την συνεργασία ε, σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας. Τα προβλήματα που ε, έθεσαν οι τρομοκρατικές απεκθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες χρήζουν απάντησης. Αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι διοργανώθηκαν δύο συναντήσεις της ΚΟΖΗ προκειμένου να, να καταρτιστούν αντιτρομοκρατικά μέτρα τα οποία συζητήθηκαν στις 29 και 30 ε, Ιανουαρίου ε, από τους αρμόδιους υπουργούς. Η ΚΟΖΗ τώρα επικεντρώνεται στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, ε, κάποια εκ των οποίων επαναλήφθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 24 Μαρτίου και ε, ο Αντιπρόεδρος ε, της ΛΥΜΠΕ, και η κυρία Γκυγιόμ παρέστη στο Συμβούλιο Υπουργών αυτών. Χρειάζεται τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια να υπάρξει συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης υπάρχει η ε, ανανεωμένη ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας για το διάστημα 2015-2020 που θα μας επιτρέψει να ε, απαντούμε σε κρίσεις καθώς αυτές θα αναδύονται. Οι συζητήσεις στην Κοζή επικεντρώνονται στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή επί Σλοβακικής και Μαλτέζικης Προεδρίας και στο επόμενο Συμβούλιο Τζάι θα παρουσιάσουμε ε, μια έκθεση για την εφαρμογή της ε, στρατηγικής αυτής. Να επισημάνω κάποιε από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και που θεωρεί η Ολλανδική Προεδρία ότι είναι απαραίτητη για την ε, ενίσχυση τη συνεργασία. Σύμφωνα λοιπόν με την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας είναι απαραίτητο να ε, καταπολεμηθεί κάθε διακίνηση ε, ανθρώπων και αποφασίσαμε να ε, επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα, ιδίως όσον, στο βαθμό που αυτό συνδέεται με την εξαγωγή εργατικού δυναμικού και την εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού, καθώς η εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού αφορά και πλήττει μια σειρά από ε, πληθυσμιακές ομάδες και κλάδους η, οδηγία, η μελέτη για την ομολογία που δημοσιεύτηκε πέρσι από την Κομισιόν ε, καταδεικνύει ότι ενδεχομένως τα ε, αδικήματα αυτά μπορούν ε, να είναι δύσκολο να αποδεικνύονται και μας λείπει πείρα. Γι' αυτό το λόγο η Ολλανδική Προεδρία αποφάσισε να καταρτήσει ένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού προκειμένου να συγκεντρωθούν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν συλλεγεί. Επίσης ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία και τον συντονισμό ε, για αυτό το ζήτημα και το θέμα θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Τζάι του Ιουνίου. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό έγκλημα, φιλοδοξία μας είναι να ε, επιτύχουμε και να δημιουργήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή δικαιοδοσία στο ζήτημα του κυβερνοεγκλήματος. Και θα συνεχίσουμε να ε, συμμετέχουμε και να ενισχύουμε και να ενθαρρύνουμε τις συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Χρειάζεται μια ε, ευρύτατη σειρά μέτρων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα αλληλοσυμπληρώνονται. για την Ολλανδική Προεδρία. Ήταν πολύ χρήσιμο το σχετικό έγγραφο που είχε εκδώσει η Λουξεμβουριανή Προεδρία. Στην Κοζή έγινε μια ανταλλαγή εμπειριών ε, σε σχέση με, τα, με τις εμπειρίες που είχαν συλλεχθεί ε, στο πλαίσιο σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση του κυβερνού εγκλήματος. Η ΚΟΖΗ λοιπόν έχει ε, καταρτήσει 30 συστάσεις που αφορούν τα κράτη-μέλη της ΕΠΟΛ, τη Europol και τον ιδιωτικό τομέα. η ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών ε, θα βοηθήσει ε, στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ενδείξεων. Επίσης, θέσαμε το ζήτημα των χρηματοοικονομικών διερευνήσεων ζητημάτων που βοηθούν στην καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος είναι να ανταλλαγεί εμπειρογνωμοσύνη και να ενισχυθεί η χρήση των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και για την βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας. Τα συμπεράσματα Συμβουλίου που αφορούν και την έχουν, έχουν καταρτιστεί και θα ε, συζητηθούν στο Συμβούλιο Τζάι του Ιουνίου η ΚΟΖΗ επίσης διοργάνωσε συζήτηση για την διοικητική προσέγγιση με στόχο την ε, αντιμετώπιση των ε, ε, ομάδων μοτοσυκλετιστών. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και διοικητικά, όχι μόνο ποινικά, και η άποψη αυτή έχει τύχει ευρύτατης αποδοχή και απήχηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να ενισχυθούν οι διοικητικέ αρχές και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για διοικητικέ υποθέσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ζητήματα αυτά ε, συζητούνται και αντιμετωπίζονται μέσω της, ε, του, του, του σημείου επαφής του, της Europol. Ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Και η ΚΟΖΗ θεωρεί ότι αυτή η διοικητική διάσταση στον ευρωπαϊκό κύκλο πολιτικής πρέπει να βελτιωθεί. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να αποτρέπουν εγκληματίες να χρησιμοποιούν ε, διοικητικές δομές και ε, να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Αυτά τα ζητήματα έχουν συζητηθεί στην Κοζή και θα εγκρεθούν στο Συμβούλιο Τζάι τον Ιούνιο. Ε, πέραν της έκθεσης που λάβατε, ε, ελπίζω να σας έδωσα μια σφαιρικότερη εικόνα για το τι κάνει η ΚΟΖΗ και σας ευχαριστούμε για την ε, ε, υποστήριξή σας στις δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άιζερμαν για τις σας πληροφορίες. Η κυρία Αναγκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Σημείωσα ότι είναι σημαντικό κι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για την κόζη. Κυρίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το τονίσατε αυτό. Ερώτηση. Σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη μας για να ανταλλάξουν πολύτιμες πληροφορίες έχουν δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες τους να συλλέξουν τις πληροφορίες, μυστικές υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή, ε, χρησιμοποιούν ανθρώπους που γνωρίζουν τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες για την πραγματοποίηση των διαφορών πράξεων, τη στρατολόγηση των μελών ή τη διοργάνωση εγκληματικών πράξεων. Έχουν εμπειρογνώμονες για τον κυβερνοχώρο. Οι οποίοι εμπειρογνώμονες μπορούν να βρουν πληροφορίες που είναι δύσκολο να βρεθούν. Και μετά, ποια είναι η σχέση με τη χρηματοδότηση αυτών των ομάδων. Αναφέρατε ότι οι οικονομικές έρευνες είναι πολύ σημαντικές. Από ό,τι βλέπω, από τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος, Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Πόρο απέχουμε από το να είμαστε αποτελεσματικοί. Κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Η ερώτησή μου λοιπόν, σε ποιο βαθμό οι τομείς αυτή; προωθούνται, κατά πόσο δημιουργούνται αμφιβολίες στην κόζη για αυτά τα θέματα σε αυτούς τους τομείς. Αναφερθήκατε στην εφαρμογή των μέτρων κατά πολεμήσεως της τρομοκρατίας. Χρειάζονται συγκεκριμένα προγράμματα από ό,τι έχουμε δει στο Κοινοβούλιο για να εμποδίσουμε τις τρομοκρατικές πράξεις, να εμποδίσουμε τη ρίζοσπαστικοποίηση να απορριζοστικοποιήσουμε ρίζοφραστικοποιημένου ανθρώπου. Τι είδου επενδύσεις κάνουν τα κράτη-μέλη για αυτό το σκοπό. Πως αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πληροφορίε στην κόζη. Γίνεται ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές και όχι αποκατάσταση και ένταξη των φυλακισμένων. Έχουμε κάνει συστάσεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας. Απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σύμφωνα με τις συστάσεις, κυρίως για τη διαμόρφωση στατικικών, σε επίπεδο κοινοτήτων κυρίως και κοινωνίας. Δεν το βλέπουμε αυτό να εφαρμόζεται. Αναφερθήκατε σε κάποιες ανησυχίες σας για το εμπόριο ανθρώπων, για την εκμετάλλευσή τους, για παράνομη εργασία. Τι κάνει η Κόζη για τη μετώπιση των ε, επισημανθέντων προβλημάτων, αυτών που επεσήμανε η Ευρωπόλ για τα 10.000 παιδιά από τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο που έφτασαν στην Ευρώπη και από αυτά τα 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί. Πώς ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται τα παιδιά αυτά για εκμετάλλευση σεξουαλική για παράνομη εργασία, για την εκμετάλλευση τους για να τους πάρουν όργανα κλπ. Είναι θέματα τα οποία τα συζητάει η Κόζη. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Ο κύριος Δίας Δεμέρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Ιζερμαν και σας ευχαριστούμε γιατί ήταν πραγματικά απαραίτητη και η επίσκεψή σας και η παρουσίαση. Και μάλιστα αυτή η δομή, αυτή η μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας είναι απαραίτητη. Ε, και είναι σημαντικό να έρχεστε πολύ πιο συχνά. Ε, γιατί δεν είναι αρκετά γνωστή αυτή η επιτροπή σα η Κόζη και το έργο τη. Μα παρουσιάσατε μία έκθεση από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή είναι η περίοδος που καλύπτει και μας παρουσιάσατε τη μεθοδολογία σας. Πριν περάσω στα υπόλοιπα σχόλια, θα ήθελα να πω ότι τρέχω ιδιαίτερο σεβασμό, ε, ε σεβασμό συγγνώμη, και ε, θεωρώ πολύ χρήσιμο το έργο σας και θεωρώ ότι ήταν απαραίτητη και αυτή η ακρόαση μαζί σας. Ε, τη μεθοδολογία φέρετε στο, θα φέρει στο τελευταίο σημείο στην αξιολόγηση επιτροπής, που κατά τη γνώμη είναι κλειδί αυτή η αξιολόγηση για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής ΚΟΖΗ για να μην είναι μια επιπλέον γραφειοκρατική διοικητική δομή ασφάλειας. 16 διαφορετικές δομές, διοικητικές δομές ασφάλειας έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ φοβάμαι, μάλλον ε, σας διαβεβαιώ ότι πολλές από αυτές τις δομές είτε αλληλοεπικαλύπτονται είτε και ε, αλλοπλέκονται και είναι καλό να γίνεται η αξιολόγηση της απειλής ε, του σοβαρού εγκλήματος και της θερμοκρατίας στην Ευρώπη. Και μας μιλήσατε και για κάποια πολυετή στρατηγικά σχέδια ε, με μεγάλη συμμετοχή των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Καλά όλα αυτά. Καλά και τα σχέδια δράσης, αλλά τέτοια σχέδια δράσης ε, κάνουν και άλλοι. Μία πλατφόρμα για τις απειλές με κέντρο τη Europol. Γνωρίζουμε τι κάνει η Europol, γιατί έρχεται πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας ενημερώσει για το έργο της. Επίσης, μας δώσατε και κάποιες πινελιές για πιο περίπλοκα θέματα. Τα έδειξε και η Αναγκόμες. Για παράδειγμα, την, το, το αίσθημα της ανασφάλειας που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη στιγμή. Επίσης, μιλήσατε για την ανησυχία της ε, Ολλανδικής Προεδρίας και το μέλημά της να αντιμετωπίσει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, αλλά και στην ε, Ευρωπόλ, οι ίδιες οι κατοχώρες στην ε, Χάγη έχουν ειδικευμένε μονάδες για το θέμα αυτό της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Φάνηκε λοιπόν, φαίνεται από όλα αυτά τα σχόλια, ότι αυτή η μόνιμη επιτροπή, η είναι αποτελεσματική δομή. Ναι ή όχι, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο μία μονάδα προβληματισμού για την ασφάλεια αλλά όχι πολλά, τίποτα, τίποτα παραπάνω και ουσιαστικά επικαλύπτεται και επικαλύπτει το έργο άλλων τέτοιων δομών ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε λοιπόν αυτή η μόνιμη επιτροπή να έχει αξιοπιστία, θα πρέπει να έρχεστε πιο συχνά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και να μα κάνετε έναν απολογισμό και παρουσίαση του έργου σα. Γιατί να μα μιλάτε για μια έκθεση που εκτείνεται από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 και να μα μιλάτε για την αξιολόγηση του 2016. Δεν ξέρω. Το άρθρο 71 έδωσε στην ΚΟΖΗ την Επιτροπή σα ο συντονισμού και συνεργασίας ε, σε ό,τι αφορά τις δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τι κάνατε σε σχέση με αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Διαδεμέρα. Δεν βλέπω να θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Έιζερμαν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας ε, κυρία Γκόμες και κύριε Δίας Δεμέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκόμες για την ανταλλαγή πληροφοριών, έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερος ε, σημαντικό στην προσπάθεια πάταξης του εγκλήματος. Και το θέμα είναι αν θα πρέπει να φροντίσουν τα κράτη-μέλη να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι και ε, επί ε, ΚΟΖΗ, επί Επιτροπής μας, αλλά και πριν, υπήρχε αυτό το ζήτημα της ε, λοιπούς ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν υπήρχε επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών για να αποτραπούν οι ε, διάφορα επεισόδια, οι, οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή να γίνει ενημέρωση. Γιατί ένα κράτο μέλο μπορεί να έχει πληροφορίε για συγκεκριμένε μορφέ εγκλήματο, αλλά δεν ενημέρωνε κατά ανάγκη και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που θα πρέπει να αναλάβει η ΚΟΖΗ, μια και μιλάμε για την αποτελεσματικότητά τη και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένω, ότι έχουμε την εντολή του Συμβουλίου να χαράξουμε έναν οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορεία για να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλους εταίρους να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανταλλάσσουν περισσότερο και καλύτερα πληροφορίες μεταξύ τους. Και τα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερος πρόθυμα και έχουν εκφράσει τη βούληση να το κάνουν. Το ίδιο και οι οργανισμοί. Στη θεωρία όμως, στην πράξη δεν είναι κάτι τόσο απλό παρά τη δεδηλωμένη βούληση όλων. Οπότε σε, σε τι βαθμό μα ρωτήσετε ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά. Θα θεσπίσουμε και αυτό το οδικό χάρτη γιατί αυτή είναι το έχουμε το Συμβούλιο. Και βέβαια εύλογα ρωτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν εφαρμόζεται και εμπράκτο. Και μάλιστα διαπιστώνουμε ότι ακόμη και αν έχουν αναλάβει δεσμεύσει τα κράτη-μέλη, δεν τι έχουν τηρήσει πάντοτε. Γιατί Και προσπαθούμε σταδιακά και προοδευτικά να ενισχύσουμε αυτή την πρακτική της ανταλλαγής των πληροφοριών. Επίσης, μας ρωτήσατε για τα ε, παιδιά. THB. Είναι κάτι που αναφέρεται, και από την Europol, γιατί έχουμε περίπου 10.000 παιδιά που κατά πάσα πιθανότητα είναι θύματα εγκληματιών και γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από εγκληματίες. Εγώ πιστεύω ότι με αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα βρούμε αυτά τα παιδιά που ίσως ακόμη και ενήλικες που είναι θύματα τέτοιας εκμετάλλευσης. Και στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας θέλουμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την ναι. ανταλλαγή των πληροφοριών και των εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα εργαλεία για να βρούμε αγνοωμένους παιδιά και ενήλικες. Και υπάρχουν και κατευθυντήρες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, και μεταξύ των θεσμικών οργάνων προσπαθούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα αυτά τα μέτρα και αυτό και θέλουμε ένα, μια πλατφόρμα εθνικών σημείων επαφής σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα του Europol, της Ευρωπόλ για τους εμπειρογνώμονες, να χρησιμοποιήσουμε και το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν και να μπορέσουμε να αναλάβουμε και αποτελεσματικέ δράσει όταν έχουμε τέτοιε καταγγελίε. Επίση, ε, γίνονται έρευνε για τη χρήση των εργαλείων και τη Interpol και για την ε, διασυνοριακή ε, ανάπτυξη μέσων προκειμένου να βρούμε τέτοιους αγνοούμενου και να γίνουν ακόμη και η κοινωνία των πολιτών τα μάτια και τα αυτιά μας για να μπορέσουμε καλύτερα να βρούμε τις αγνώμενες. Επίσης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, γραμμές τηλεφωνικές για καταγγελίες και θέλουμε με την ανάμεξη φυσικά των πολιτών να εκφράσουμε την προσήλωσή μας στην τήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων και φυσικά να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε των πολιτών αλλά και τι ιδιαιτερότητε μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Και μάλιστα στι 25 Μαου την ημέρα του αγνοούμενου παιδιού θα οργανώσουμε και μία ειδική διάσκεψη για τους αγνοωμένους στο Άμστερνταμ και θα αξιοποιήσουμε και το έργο αυτής της διάλεξης για να ε, βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας. Ο κύριος Ντίας Μέρα μας ρώτησε αν είμαστε μια πραγματικά αποτελεσματική μόνιμη επιτροπή, είμαστε απλώς ένα επιπλέον διοικητικό σώμα. Αν δείτε την ιστορία της μόνιμης αυτής επιτροπής ΚΟΖΗ, διαπιστώνεται ότι προκύπτει από την συνθήκη της Λισαβόνας και στόχο έχει την πρόθεση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή αυτή από μόνη της ασκεί επιχειρησιακές δραστηριότητες. Πάντως, ε, μετά από λιγόμενη εμπειρία στην Προεδρία της ΚΟΖΗ, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς όπως την Ευρωπόλ, τη Eurojust, τη Frontex, να συνεργάζονται σε αυτόν τον κύκλο της πολιτικής. Και φυσικά υπάρχει και εδώ κάποια γενής γραφειοκρατία. Αλλά σε τελική ανάλυση, όταν έχουμε συνεργασία με 28 χώρες και με τόσου διαφορετικούς οργανισμούς και δομές, χρειαζόμαστε και κάποια μορφή οργάνωσης, μια οργανωτική δομή. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι η ΚΟΖΗ βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τη. Και μα ζητήσατε να ερχόμαστε πιο συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω, πολύ ευχαρίστω να ξαναέρθω. Ε, και θα μεταβιβάσω αυτή την επιθυμία σας και στην ε, επόμενη Προεδρία της ΚΟΖΗ. Γιατί έχουμε κοινό ζητούμενο να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις. Αναφερθήκατε και στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει μονάδα αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος στη Europol, στην Ευρωπόλ. Και ε, κάποιες χαρισμένοι έχουν αντίστοιχες μονάδες πάταξης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Και εμείς στην Ολλανδική Προεδρία προσπαθούμε να πάμε λίγο ακόμη πιο μακριά. Και όταν έχουμε απώλεια ε, εντοπισμού έλλειψη της θέσης, ε, ε, τα μέσα επιβολή του νόμου αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας διαφορά των συστημάτων. Και δοκιμάσαμε πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργηθεί μια νέα επί, περιοχή της τρομοκρατίας, ένας άλλος χώρος τρομοκρατίας, ο κυβερνοχώρος, που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία με... και που δεν καλύπτεται μέχρι στιγμής από τα υπάρχοντα συστήματα. Μάλιστα είχαμε κοινέ ε, ημερίδες δράσεις για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και διαπιστώσαμε ότι οι διάφορες αρχές θεωρούν αναγκαίο να βρεθούν κάποιες ε, ε, λύσεις που αφορούν τη δικαιοδοσία, την ε, απώλεια χώρου και ούτω καθεξής. Και αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Απώλεια θέση, συγγνώμη. Αυτά και νομίζω ότι απάντησε σε ερωτήσεις. Η κυρία Γκόμε, συμπληρωματική. Συγγνώμη. Θα ήθελα να απαντήσετε και στο ερώτημα για τις ε, προσπάθειες πολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Η ΚΟΖΗ έχει ε, επαρκή στελέχωση στα κράτη-μέλη προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες ε, ενέργειες και ε, βλέπω, βλέπω ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι ίδιες οι τράπεζες λειτουργούν ως μηχανισμός ξεπλήματος χρήσης. Μήπως θα έπρεπε και αυτά τα ζητήματα που ανέδειξαν τα Panama Papers να τα να, να τα εξετάσουμε πιο σοβαρά. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα που χρησιμοποιείται και αξιοποιεί τα, τα δικά μας συστήματα. Να απαντήσετε επίσης, παρακαλώ, αν ε, αν έχετε αναλάβει δράση για την αποτροπή και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και αν κάτι τέτοιο υπάρχει στην ατζέντα, στο θεματολόγιο που συζητάει η Κοζή. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν απάντησα στο ζήτημα της πρόληψης. Ναι, αποτελούν τμήμα των ε, προτεραιοτήτων που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο με στόχο την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και την πρόληψη της τρομοκρατίας. Και αυτό υπάρχει βεβαίως ως θέμα και στο πρόγραμμα της ΚΟΖΗ. Επίσης, ρωτήσατε ποιε είναι οι επενδύσεις των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Ε, η ΚΟΖΗ δεν συζητά αυτά τα θέματα. Δεν είναι ένα ζήτημα που έχουμε προβλέψει εμείς. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στο Συμβούλιο για να συζητηθούν οι δυνατότητες στον τομέα της πρόληψης. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό δεν αφορά τόσο πολύ την ε, επιχειρησιακή συνεργασία. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλά στην ε, ατζέντα μας, αλλά έχετε δίκιο, συμφωνώ και εγώ, ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Ε, όχι μόνο δηλαδή στην καταπολέμηση, αλλά και την πρόληψη της τρομοκρατίας. Όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικο χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και αναφερθήκατε και στα Panama Papers, ε, θα γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει καταρτιστεί πλέον και η Κομισιόν θα υποβάλει και μια πρόταση σύντομα σχετικά με την καταπολέμηση της ε, ε, νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό ωστόσο αφορά το υπόβαθρο για το έργο της ΚΟΖΗ Φυσικά το ξέπλυμα, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, συνδέεται με, την, ε, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά ε, γνωρίζετε ότι και σε επίπεδο κρατών μελών είναι ένα θέμα δύσκολο και έτσι είμαστε εν αναμονή της σχετικής πρότασης που θα, που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Ίζερμαν, λέει Πρόεδρος, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και στο μέλλον το έργο της ΚΟΖΗ. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες σας, τις πολύ σημαντικές εργασίες σας. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ναβαρέτε, που είναι επικεφαλής του νεοπαγού Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας της Europol και καθώς η ε, παρέμβαση του είχε ε, προγραμματιστεί να γίνει στις 5 παρατέταρτο έχουμε περίπου 20 λεπτά, 25 περίπου ε, για να περιμένουμε Αναστέλω λοιπόν την συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στις 16.45 όταν και θα καταφτάσει εδώ ο κύριος Ναβαρέτε, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Κατολέμηση της Θερμοκρατίας. Uh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με την απογευματινή μας συνεδρίαση. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ναβαρέτε, που είναι επικεφαλής του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καποτελέμηση της Τρομοκρατίας στην Europol. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο κύριος Ναβαρέτε θα μας παρουσιάσει την έκθεση για την ε, κατάσταση τρομοκρατίας 2016 και την πρόσφατη δημοσίευση με τίτλο «Αλλαγές στο μόντους operandi των τρομοκρατικών πεθέσεων του Ισλαμικού κράτους». Σας δίνω το λόγο. Αμέσως, κύριε Ναβαρέτε, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση με τους βουλευτές. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κυρίως ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Είμαι ενώπιόν σας για να αναφερθώ σε κάποια από τα πορίσματα της Europol όσον αφορά τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και να επενέσω κάποιες κοινέ προσπάθειες που ήδη έχουν γίνει και αυτές που ήδη απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε τις τρομοκρατικές απειλές και να κάνω συστάσεις. Κάθε χρόνο, που ξέρετε, η Europol εκπονεί αναδρομική ανάλυση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Η, η έκθεση TSAT, της πράξης και της τάσης τρομοκρατικών αριών. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας Ευρωπόλ και κρατών μελών και συνεργασία με την Eurojust, INSEM και συνεργασία και με τρίτες χώρες ε, συμμετέχουν στην προσπάθεια. Είναι μια πολύ καλή εικόνα της τρομοκρατικής απειλής και πώς αλλάζει αυτή. Κάτι που επηρεάζει βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση, η TISA του 2016, θα είναι διαθέσιμη μόνο στο διαδίκτυο σε μερικές εβδομάδες. Παρόλα αυτά όμως δράτωμα της ευκαιρίας να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα βασικά πορίσματα της εκθέσεως. Θα συνδυάσω τη σημερινή μου παρουσίαση με τα βασικά συμπεράσματα της TSAT 2016 και τις διάφορες συστάσεις που ετοιμάσαμε πριν από τις επιθέσεις του Νευρίου του 2015 Δηλαδή πώς άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της το Ισλαμικό κράτος, ε, τον τρόπο λειτουργίας του το Ισλαμικό κράτος και τον τρόπο επιθέσεων. Και στο συμπροματικό κείμενο της ΤΙΣΑ 2016 αναφερόμαστε περαιτέρω στην αλλαγή του Μόντου Operandi. Και πώ ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρομοκρατία είναι ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί. Θα παρουσιάσω κάποιο από τι πρωτοβουλίε τη Europol. Θέλουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία, θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Βλέπετε τώρα στην οθόνη, στις διαφάνειες, τα βασικά πορίσματα της T-SAT 2016. Το 2015, 151 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 360 ανθρώπους τραυματίστηκαν σαν αποτέλεσμα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το συγκρίνουμε αυτό με τα στοιχεία του 2014 βλέπουμε ότι πριν από ένα χρόνο τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συγκρίση με 151 ανθρώπους που σκοτώθηκαν το 2015. Πέραν αυτού, 60 πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως σκοτώθηκαν σε διάφορες επιθέσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως στην την Ισία. Ε, 211 ε, επιθέσεις απέτυχαν ή εμποδίστηκαν ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση των αστυνομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας ε, ήταν κάτι που τονίστηκε ιδιαίτερα, Κατεβλάθησαν προσπάθειες τεράστιες. 1057 άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πράξεις που σχετιζόταν με τρομοκρατία. Το 2015 ήταν ένα έτος όπου έγιναν πολλές δίκες σχετικά με τις τρομοκρατικές πράξεις. 513 άτομα κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία ε, και ολοκληρώθηκαν οι, οι συγγνώμη, υποθέσεις αυτές το 2015, δικαιρεώθηκαν. Επόμενη διαφάνεια. Τώρα, Πάμε σε συγκεκριμένους ε, τομείς των διαφόρων απειλών που εστρέφονται κατά της Ευρωπαϊκής από 150 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τους τρομοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 150 από αυτούς ανθρώπους σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές, τζιχαντιστικές ομάδες εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 150 άνθρωποι λοιπόν σκοτώθηκαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών. Έχουμε σημαντική αύξηση του αριθμού τζιχαντιστικών επιθέσεων από 4 το 2014 φτάσαμε στις 17 επιθέσεις το 2015. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι θύματα είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συμμετείχαν στη συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους θεωρούνται τα κράτη-μέλη από τις ομοκρατικές ομάδες σαν θεμητοί ε, στόχοι των ομάδων. Όπως αναφέρθηκα και αρχικά σε αυτό το θέμα, όπως σας είπα στην αρχή, οι αστυνομικέ δυνάμεις και οι δυνάμεις του νόμου ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες αντιμετωπίσεως του φαινομένου, ήταν σχερή αντίδραση. Από 395 άτομα που συνελήφθησαν το 2014 φτάσαμε στα 667 άτομα του 2015. Λοιπόν, οι τρομοκρατικές ομάδες είναι έτοιμες να επιτεθούν. Ε, μάλλον οι τρομοκρατικές ομάδες ήταν εντόπιες κυρίως, αλλά έχουν σχέσεις με το Ισλαμικό κράτος, το ούτως αποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος. Η επόμενη διαφάνεια. η βασική ανησυχία των κρατών μελών, ανησυχίες που αναφέρονται στην έκθεση της ΣΑΤ του 2016, είναι η τζιχαντιστική τρομοκρατία και το φαινόμενο των ε, ξένων μαχητών ε, που ταξιδεύουν, πηγαίνουν στις ε, περιοχές με συγκρούσεις χώρες των συγκρούσεων και επιστρέφουν. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε τον ορισμό της τζιχαδιστικής τρομοκρατίας για να χαρακτηρίσουμε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο αριθμός των συλλήψεων τζιχαντιστών ε, αυξήθηκε το 2015 εν συγκρίση με το 2014. Αυτό δείχνει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται σε όλη την Ευρώπη για την καταπολέμηση αυτού του είδους της ε, τρομοκρατίας. Πάμε τώρα στο ιστορικό των τζιχαντιστών. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εικόνα τζιχαντιστού. Η μεγάλη πλειοψηφία των στατολογηθέντων έχουν εγκληματικό παρελθόν. Από μικρό έγκλημα και σε... φτάνουμε στα πιο σοβαρά εγκλήματα στο παρελθόν αυτών των ατόμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες χώρες, σημαντικό ποσοστό των ξένων μαχητών ε, διαπιστώθηκε ότι είχαν ε, ψυχικά προβλήματα η εκπαίδευση είναι σημαντική συνιστόσα της τρομοκρατίας της τζιχαντιστικής. Κάποιοι εκπαιδεύτηκαν στη Συρία για να διαπράξουν επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη τυπολογία του τζιχαντιστή τρομοκράτη είναι ο ξένος μαχητής που ανεξάρτητα οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτός όταν επιστρέψει από την Ισλαμιστική χώρα στην Ευρώπη γίνεται κάποια εκπαίδευση από ό,τι ξέρουμε εντός των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν το έχουμε παλιθεύσει κατά πόσο ισχύει. Οι τρομοκράτες εκπαιδεύονται κυρίως στη χρήση πυροβόλων όπλων και κρυκτικών. Η τελευταία κατηγορία ε, είναι απειλή, μεγάλη απειλή για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Εν γέννη, είναι πλήρως εκπαιδευμένοι αυτοί και είναι απρόβλεπτη. Άρα δύσκολο να εμποδίσουμε μια τρομοκρατική ε, επίθεση από αυτούς τους ανθρώπους που είναι δραστηριοποιημένοι επί μακρόν χρονικό διάστημα. Και είναι μεγάλη απειλή για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτού, αρκετοί Ευρωπαίοι τζιχαντιστές έχουν πολύ σημαντική θέση στο ούτως αποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος και κρατούν επαφές με τρομοκρατικά δίκτυα των ε, χωρών καταγωγής. Όσον αφορά τους στόχους, φαίνεται ότι οι τρομοκράτες προτιμούν τους μαλακούς αποκαλούμενους στόχους. Περισσότερο επιτίθεται παρά κατά των πιο σοβαρών υποδομών, σκληρών στόχων όπως αποκαλούνται, όπως είναι αστυνομικές μονάδες, αστυνομικές αστυνομικά τμήματα, διάφορε θετικέ εγκαταστάσει κλπ. Παραμένει όμω η δυνατότητα να επιταθούν κατά αυτών των σκληρών αποκαλούμενων στόχων. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά του ε, νασιοναλιστέ, ε, του εθνικιστέ και του αποσχιστέ τρομοκράτε. Οι επιθέσει από αυτέ τι ομάδε μειώνονται. Από 65 φτάσαμε σε 65 του 2015 επιθέσει από εθνικιστικέ ομάδε. Υπήρξε έντονη αντίδραση αστυνομικών δυνάμεων κατά αυτών των ομάδων. 168 άτομα συνελήφθησαν για δικήματα που σχετίζονται με αποσχιστική τρομοκρατία, εθνικιστική τρομοκρατία, ε, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2014. Τα περισσότερα γεγονότα τα είχαμε στην Γαλλία και την Ισπανία. στην αστυνομική υπηρεσία ε, της Βορείου Ιρλανδίας, PSNI, είναι βασικός στόχος των αποσχιστικών ρεπουμπλικανικών ομάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε δει κίνδυνο ε, ε βίες αντιπαράθεσης μεταξύ αποσχιστικών δυνάμεων υπέρ των Κούρδων και τουρκικών εθνικιστικών ε, δυνάμεων στην, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μετά πάμε σε άλλο τομέα, σε άλλη διαφάνεια επιθέσεις από αποσχιστές και αριστερούς ε, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα μετά το 2006. Είχαμε 67 άτομα που συνελήφθησαν σε 6 κράτη-μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτές τις επιθέσεις είχαμε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το βασικό όπλο που χρησιμοποιούν αυτές οι ομάδες. Οι ριζοσπαστικές ομάδες μαρξιστιών, λενινιστών κυρίως ασχολούνται με προπαγάνδα και στατολόγηση αν θέλετε μελών αλλά δεν έχουν προβεί σε κάποιες ε, βίες πράξεις μέχρι τώρα. Τώρα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, διαδίδεται ένα συνέστημα κατά των μεταναστών και κατά του Ισλάμ και ο εξτρεμισμός της δεξιάς έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο, αυξάνεται η αστηριότητα αυτής της πτέρυγας σε κάτι μεσολογικής ενώσεως. Δεν είχαμε επιθέσεις το 2014, καμία, μηδέν. Τώρα έχουμε 9 επιθέσεις που έλαβαν χώρα το 2015 που σχετίζονται με ακροδεξιές ομάδες και τρομοκρατία ακροδεξιών ομάδων. Λοιπόν, οι συλλήψεις των ακροδεξιών αυξήθησαν από 34 άτομα το 2014 Μάλλον μειώθηκαν εδώ. Μειώθηκαν. Φτάσαμε στι 11 το 2015, με συγχωρείτε. Πάμε στην τελευταία διαφάνεια εδώ, στην επόμενη διαφάνεια. Στις επιθέσεις που έγιναν στο Παρίσι το Νοέμβριο, αλλά και φέτος εδώ, στην καρδιά των Βρυξελών στις Βρυξέλλες, είδαμε ότι οι τζιχαντιστές τρομοκράτες χρησιμοποιούν νέες τακτικές νέες τεχνικές χρησιμοποιούν ε, εκρηκτικά. Ήταν η πρώτη φορά που το Νοέμβριο του 2015 χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός εκρηκτικών και όπλων πυροβόλων για να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν ανθρώπους στο Παρίσι. Τα οικιακά εκρηκτικά, αυτά που κατασκευάζονται στο σπίτι, από, τα κατασκευάζουν οι ίδιοι οι τρομοκράτες, είναι η πιο διαδεδομένη εκρηκτική ουσία που χρησιμοποιείται. Και έχουμε κάποιε πληροφορίε που μα δόθηκαν από το Κατημέλιο ότι ότι τρομοκρατικέ ομάδε προσπάθησαν να δημιουργήσουν ε, ε, ε διάφορες αποθήκες ε, ε, με εκρηκτικά και διάφορες ουσίες, πρόδρομες ουσίες για την κατασκευή εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις με εκρηκτικά μεγάλη κλίμακας. Τώρα, εργαστήρια για την παραγωγή χημικών ουσιών. Ε, μάλλον η εργοστάσια χημικών ουσιών είναι ευάλωτοι στόχοι. Χρησιμοποιούν όμω παραδοσιακά εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα οι τρομοκράτες. Είναι πιο εύκολα διαθέσιμα. Είναι πιο απλά μέσα και είναι και αποτελεσματικά. Αντί να χρησιμοποιήσουν βιολογικές ουσίες και άλλε ουσίε. Και τώρα πάμε σε άλλη διάσταση. κατάχρηση χρήση μάλλον του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων από πλευρά τρομοκρατών. Το διαδίκτυο και των σχετικών υπηρεσιών και των υποδομών αυτών είναι και μέσα επίθεσης αλλά και στόχος. Το 2015 αυξήθηκε η χρήση και η κατάχρηση της ανωνυμίας των υπηρεσιών κρυπτογράφησης και των διαφόρων εργαλείων για να μπορεί να αποκρύπτεται η γεωγραφική τοποθεσία, να προστατεύονται τα στοιχεία και επικοινωνίες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Άρα είναι πιο δύσκολη η παρακολούθηση από πλευράς αστυνομίας. Και είναι και πιο δύσκολος ο εντοπισμός των παρανόμων ε, οικονομικών ε, συναλλαγών με αυτόν τον τρόπο. Γιατί καλύπτονται οι δραστηριότητε τους. Αυτά είναι τα βασικά απορίσματα της εκθέσεως του 2016. σε σύγκριση με το 2015 βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η απειλή αλλάζει. Κυρίως όσον αφορά τις τζιχαντιστικές ομάδες και τις σχέσεις που έχουν αυτές με το Ισλαμικό κράτος. Είδαμε και τη δράση των αστυνομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας για την αμετώπιση του κινδύνου. Να σας πω τώρα ποιες ήταν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κυρίως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου που δημιουργήθηκε το, αρμόδιο κέντρο στη Europol για την καταπολέμηση του φαινόμενου. Τα τραγικά γεγονότα του τελευταίου μήνα του 2015 αλλά και των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους επιβεβαίωσαν ότι η τζιγαντιστική τρομοκρατία είναι η μέγιστη απειλή για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, 30 άτομα σκοτώθηκαν εδώ στις Βρυξέλλες το 2016 αλλά και πολλοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σκοτώθηκαν από τρομοκράτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη και στην ακτή του Ελεφαντοστού. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη ανέπτυξε μια ισχυρή πολιτική απάντηση για αντιμετώπιση την αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή. Επιτέλους ολοκληρώθηκαν νομοθετήματα στα πλαίσια της θεσμικής ε, συνεργασίας. Η Europol ήταν βασικός φορέας της προσπάθειας. Για να βρούμε απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της τρομοκρατικής απειλής. Το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, μας στήριξαν στη διαδικασία. Δράτω με να σε ευχαριστήσω εκ νέου για την υποστήριξή σας. Για την εφαρμογή ενός νέου κανονισμού της για τη Europol και για τη διάθεση πραγματικών πόρων για να δημιουργηθεί το νέο κέντρο καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας στην Europol. Έτσι θα γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η αντίδραση της Europol μετά σε επιθέσεις στο Παρίσι ήταν άμεσες. Είμαστε στενή επαφή με τη Γαλλία μετά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι δημιούργησαν μια ομάδα ε, για κατεπίγουσας ανταπόκρισης για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους που υπέφεραν τις επιθέσεις. Περίπου 60 ε, αξιωματικούς είχαμε που δούλευαν 24 ώστε 24 ώρα για να στηρίξουμε τους ε, Γάλλους και δώσαμε αμέσω στη Γαλλία υποστήριξη όσον αφορά οικονομικές συναλλαγές. Σε 6 ώρες δώσαν πληροφορίες για οικονομικές συναλλαγές, 6 ώρες μετά την επίθεση και περισσότερες πληροφορίες δόθηκαν για επιθέσεις κατά στον κυβερνοχώρο και ε, επίσης έγινε άμεση ανταλλαγή και διαβίβαση πληροφοριών πλευράς Europol προς τη Γαλλία. Δημιουργήσαμε μόνιμη ομάδα, μετά μερικές ομάδες, για να στηρίξουμε τους Γάλλους συναδέλφους και τους Βέλγους συναδέλφους. Όταν βρήκαμε ότι υπήρχε και σχέση με το Βέλγιο, για να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, όλους τους πόρους, για να υποστηρίξουμε τη Γαλλία και το Βέλγιο και για να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Ξέραμε ότι υπέφεραν δύο κράτη-μέλη, αλλά έπρεπε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες που είχαμε σε διάσταση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για να, για να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γιατί η απειλή είχε πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Θέλαμε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και είχαμε, δημιουργήσαμε ομάδα κρούσης με το όνομα Φρατερνιτέ. το σκοπό μαζί με εμπειρογνώμονες και αξιωματικούς συνδέσμου, ε, συνδέσμους της Γαλλίας και του Βελγίου προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τις δύο χώρες με τις επιθέσεις. Η Φρατερνιτέ υποστηρίζει τη Γαλλία και το Βέλγιο μετά τις επιθέσεις που υπέστησαν. Επίσης βρήκαμε και σχέσεις που υπήρχαν με άλλα κρατημέλη και έχουν συνδεθεί και άλλα κρατημέλη ε, με αυτή την ομάδα κρούσης. Το, κέντρο, το Αντιδημοκρατικό Κέντρο, το Ευρωπαϊκό, στη Europol, βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα και στις δυνατότητες που έχουμε. Ξεκίνησε εργασίες επισήμως τον Ιανουάριο του 2016. Είναι μια βάση που συνδυάζει διάφορα εργαλεία. Το αντιτρομοκρατικό αυτό κέντρο ε, κάτω από μία στέγη ε, συγκαταλέγουμε διάφορες δυνατότητες για την μετώπιση τρομοκρατικής απειλής. Το κέντρο αυτό αντιπροσωπεύει τη γενική φιλοσοφία και στρατηγική της Europol. Έχουμε ένα κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών, δίνουμε επιχειρησιακή ανάλυση ε, στα διάφορα κάτι μέλη για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις Εξετάζουμε πώ χρηματοδοτούνται, πώ συλλέγουν όπλα, πώ διαβιβάζουν στο διαδίκτυο του προπαγάνδα οι τρομοκράτε μέσω του κέντρου αυτού. Και έχουμε μια καινοτόμα βάση για να οργανώνουμε τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να καταπολεμούμε καλύτερα την τρομοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Ένας από τους πυλώνε του κέντρου είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Περισσότερη ανταλλαγή ε, πληροφοριών αλλά και προστατούμε με τη χρήση της αλλά και την αξιοποίηση της βασικού παίκτη να καθοδηγήσουμε τις βασικές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες. Επίσης, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να στείλουν στην Europol συγκεκριμένους ε, αξιωματικούς συνδέσμους ε, με επιχειρησιακά σχέδια που βρίσκονται στο βασικό θεματολόγιο, βασικές προτεραιότητες των αρμόδιων αρχών και χρησιμοποιούμε και του πόρους του Ευρωπόλ για να το στηρίξουμε. Και μάλιστα ε, πρόκειται για ενέργειες ε, οποίε οποίες ε, εφαρμόζουν τα κρατη με την υποστήριξη της Europol και θα πρέπει ε, αυτές οι ενέργειες να είναι μετρήσιμες, αναθεωρήσιμες και φυσικά εφικτέ. να αποφέρουν καρπού κράτη-μέλη έστειλαν αξιωματικού συνδέσμου για να συνεργαστούμε με την Europol και να μπορέσουμε να του βοηθήσουμε στην ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρε και η Γερμανία έχουν ήδη στείλει τέτοιου αξιωματικού συνδέσμου. Αλλά και άλλε χώρε έχουν αναγγείλει την αποστολή εμπειρογνωμόνων στο αντιτρομοκρατικό μα κέντρο για να συντονίσουμε καλύτερα ενέργειες που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόσφορο ε, κλίμα για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Και μάλιστα, ε, ειδικά για, την, ε, για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, έχουμε το CNACT στο σύστημά μας. Όλοι πια ε, έχουν συνδεθεί σε αυτό το σύστημα για ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα για τον αντιτρομοκρατικό μας αγώνα. Και μέχρι στιγμή τα κράτη-μέλη, αλλά και τρίτες χώρες, 43 αρμόδιες αρχές, ε, αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί σε αυτό το σύστημα, CTCNR προς το παρόν. Και μάλιστα το σύστημα θα γίνει εμπιστευτικό, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα διαβαθμισμένε. διαβαθμισμένες. Μέχρι στιγμής έχει αρχίσει και λειτουργεί το σύστημα. Η ανάλυση των πληροφοριών είναι βασικό καθήκον και έργο της Europol. Η επιτυχία του αντιτρομοκρατικού μας κέντρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Europol να διευκολύνει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και κάτι που βελτιώθηκε μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη ε, με μεγαλύτερη προθυμία πια χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της Europol, γιατί αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ή μάλλον τη ραχοκοκαλιά της Europol αυτό το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και τροφοδοτείται άμεσα από τα κράτη-μέλη. Εμείς απλώς συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες στο σύστημα πληροφοριών της Europol και ε, εντάσσουμε πληροφορίες και από, τρίτα μέρη, από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα για το φαινόμενο των ξένων μαχητών, τα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες έχουν εντοπίσει 18 ε, τέτοιους ε, στο σύστημα μέχρι τα τέλη του 2014, ενώ έχουμε περάσει τώρα στους 4.000. Από 18 το 2014 έχουμε εντοπίσει 4.000 ξένους μαθητές σήμερα. Επίσης, από από την σύσταση του εστιακού σημείου για τα πυροβόλα όπλα το Σεπτέμβριο του 2015 έχουμε πολλές πληροφορίες και έχουν ξεκινήσει 600 και έρευνες για τα θέματα αυτά, για τα πυροβόλα όπλα και την κατοχή τους. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε το σύνδεσμο οργανωμένων εγκλήματος και τρομοκρατίας. Και όπως είπα και στην αρχή, έχουμε διαπιστώσει ότι οι περισσότερες η περισσότερη αυτούργη, η φυσική αυτούργη τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια είχαν ε, εγκληματικό παρελθόν. Το κέντρο μας καταπολέμησης της τρομοκρατίας ε, ενισχύει και τις ε, δυνατότητες συγκέντρωσης οικονομικών πληροφοριών. Και μάλιστα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις η Γαλλία Μα ζήτησε πρώτα απ' όλα πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα. Και μάλιστα με τη χρήση του προγράμματος ε, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορέσαμε πέρυσι να δώσουμε πάνω από 2.700 στοιχεία στα κράτη-μέλη ε, οικονομικού χαρακτήρα. Μάλιστα έχουμε και ένα ε, δίκτυο οικονομικών πληροφοριών στην Europol ενισχύοντας την προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία χρησιμοποιώντας ε, οικονομικές πληροφορίες για τα κυκλώματα αυτά. Οπότε, καλή βέβαια η αντιμετώπιση και η ελαχιστοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά η πρόληψη είναι ακόμη καλύτερη και το κέντρο μας ε, διαδραματίζει ρόλο και στην πρόληψη με τις online έρευνες, γιατί οι τρομοκρατικές ε, οργανώσεις έχουν αντιληφθεί τη λειτουργία των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα χρησιμοποιούν ε, στις προπαγάνδες τους για τη στρατολόγηση οπαδών, για τη διευκόλυνση της σπαστικοποίησης, την προώθηση τρομοκρατικών ενεργειών και την εξήμνηση των υποδαβλισμών του εξτρεμισμού, αλλά και για την συγκέντρωση κονδυλίων. Πάνω από 50.000 λογαριασμοί Twitter είχαν χρησιμοποιηθεί από το Ισλαμικό κράτος ε, και εκατομμύρια tweet ε, ε, καθημερινά γίνονται για το θέμα αυτό. Είναι ύπουλη αυτή η απειλή. Μάλιστα η Twitter εντόπισε 125 ισλαμιστικούς, τζεχαντιστικούς λογαριασμούς από Γι' αυτό και καλό είναι να επικεντρωθούμε στην πρόληψη που θα είναι και βασικό θεμέλιο του αντιτρομοκρατικού μας αγώνα. Και γι' αυτό έχουμε και την ε, μονάδα ε, ψηφιακού περιεχομένου, αναφορά ψηφιακού περιεχομένου που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, βρισκόταν σε πειραματική φάση και εντρεώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Να σα δώσω κάποια στοιχεία. Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Μάλιστα έχουμε εντοπίσει πάρα από 17.000 ε, ε, ύποπτο περιεχόμενο ψηφιακό, αυτή η μονάδα αναφοράς ψηφιακού περιεχομένου. Και επιτυχής ε, αναφορά ψηφιακού περιεχομένου αφορά το 90% των καταγγελιών που έγιναν από την μονάδα αυτή στο κέντρο αντιτρομοκρατίας της Ευρωπόλ. Και τέλος, λίγα λόγια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ε, με τις τελευταίες ε, επιθέσεις, ε, αντιπιστώσαμε ότι ε, οι τρομοκράτες έχουν βελτιώσει το συντονισμό τους από ό,τι στο παρελθόν και χρησιμοποιούν όχι μόνο εκρηκτικά αλλά και πυροβολά όπλα. Χρησιμοποιούν όχι μόνο ε, μαχητές που έχουν επιστρέψει και τρομοκράτες που έχουν επανέλθει από εμπόλεμες ζώνες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά ε, παροτρύνουν και ντόπιου ζυχαντιστέ να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους και να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απειλή κινείται με ραγδαίους ρυθμούς, αναπτύσσεται γρήγορα και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, διασύνδεση ε, ποινικών εγκληματιών και τρομοκρατών. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Επίσης, ε, οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προπαγάνδα τους. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην ε, ε, εξάρθρωση αυτής της προπαγάνδας και ένα τμήμα αυτού του ρόλου το αναλαμβάνει η Ευρωπόλ και το κέντρο μας. Τώρα, συγκεκριμένες έρευνες. Φυσικά βοηθήσαμε τη Γαλλία και το Βέλγιο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε αυτές τις χώρες και να λαμβάνουμε πληροφορίες από τις υπόλοιπες χώρες προκειμένου να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Πρόσφατα η Ευρωπόλ έχει γίνει σημαντικός παίκτη της αντιτρομοκρατίας και χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κέντρο μας και στην πολιτική όθηση που λάβαμε ε, τα προηγούμενα χρόνια, 2014 και 2015, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτά και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ναβαρέτε και ευχαριστούμε για την ενδελεχή και μεστή παρουσίαση που μας κάνατε. Παρακαλώ τώρα οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχω ο κύριο Χάλα Άχολε. Έχω κάποιες, πληροφο... Έχω κάποιες ερωτήσεις για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Ε, δεν μας δώσετε στοιχεία για τις επιθέσεις ε, από αναρχικούς και αριστερούς. Γιατί αναφερθήκατε σε σχέδιο και κρυπτικούς μηχανισμούς που είναι ε, το μέσο που προτιμούν τέτοιες ομάδες για τις επιθέσεις τους ε, που είτε διαπράττουν είτε επιχειρούν και ματαιώνονται. Επίσης, με ενδιαφέρει η φύση της αριστερής τρομοκρατίας ε, και αναρχικής, ε, ποιο είναι, τι βρίσκεται στο στόχαστρο, άλλες εξτρεμιστικές ομάδες ή απλοί άνθρωποι. Και υπάρχουν θύματα τέτοιων ε, ενεργειών, ιδιαίτερα στα κρατη έχουμε περισσότερα θύματα σε ορισμένα από ό,τι σε άλλα. Και μιλώ για την τρομοκρατία των αριστερών ομάδων. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα στο έργο του κέντρου και ευχαριστώ ε, έναν κορυφαίο επαγγελματία στον κλάδο της αντιτρομοκρατίας ε, και σας ευχαριστώ που ασχολείστε και μεριμνάτε για την ασφάλεια των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Ε, μιλήσατε για τα θέματα που μας απασχόλησαν περισσότερο τους τελευταίους μήνες και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ήταν τα θέματα που μας προβλημάτισαν κατεξοχήν και χαίρομαι που μας δώσατε με απλά λόγια και σε πρώτη παρουσίαση τα συμπεράσματα της ΤΕΣΑΤ και του νέου σύστατου αυτού κέντρου καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και μας είπατε τι νομικές και νομοθετικές δυσκολίες που είχαμε για την ε, μονάδα αναφοράς ψηφιακού περιεχομένου. Γιατί πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήθελαν να διαχωρίσουν την μονάδα αυτή από την Europol. Τελικά καταφέραμε να την περιλάβουμε και αυτήν την ομάδα, την IRU, την ομάδα αναφοράς ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρωπόλ. Και φαντάζομαι θα γνωρίζετε ότι είχαμε εκτενέστατες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σφοδρές συζητήσεις για το θέμα αυτό, για να στηρίξουμε και να δώσουμε και νομική βάση σε αυτή τη μονάδα αναφοράς ψηφιακού περιεχομένου για να εξουδετερώσουμε την τζιχαντιστική προπαγάνδα στο διαδίκτυο. Και από αυτή την άποψη, εσείς είστε, όπως σας είπα, κορυφαίος εμπειρογνώμονας στα θέματα αυτά και είστε και ο διευθυντής αυτού του κέντρου αντιτρομοκρατίας. Μετά τις εξηγήσεις που δώσατε στην ομάδα εργασίας για τον κανονισμό για τη Europol, θα ήθελα να μας πείτε γιατί η ταχύτητα ε, και η ανθεκτικότητα ε, είναι στοιχεία που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και μόνο η Ευρωπόλ μπορεί να το κάνει και πολύ καλύτερα από ό,τι τα μεμονωμένα κρατημέλη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, μιλήσατε για τα χαρακτηριστικά και την εκπαίδευση των ε, τζιχαντιστών και τρομοκρατών. Σε πολλά ε, μέσα ενημέρωσης ακούμε για το ρόλο της γυναίκας της διχαντίστριας, πώς εκπαιδεύονται και πώς ετοιμάζονται οι γυναίκες της διχαντίστριας. Γιατί δεν είναι εύκολο να ενταπιστούν για την έγκαιρη προειδοποίηση. Τουλάχιστον δεν εντοπίζονται τόσο εύκολα όσο οι αντίστοιχοι, οι αντίστοιχοι άνδρες διχαντιστές. Έχει βάση αυτή η πληροφορία. Είναι πραγματικά ε, πραγματική απειλή αυτή η θανατηφόρα συμμετοχή αυτών των τζεχατιστριών που ακούσαμε ότι πέντε στη Συρία, αλλά πολύ πιθανό να γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σα, ε, τι ειδικευμένε πληροφορίε που μα δώσατε και σα ευχαριστώ και πάλι θερμά ε, για την προσήλωσή σα στην ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Κύριε Γκόμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ναβαρέτε, για την παρουσίασή σας. Σημειώνω ότι μας δώσατε στατιστικά στοιχεία για το 2015. Δυστυχώς βεβαίως οι αριθμοί αυξάνονται το 2016. Αλλά είναι σημαντικό να το θεωρήσουμε όλο αυτό και στο πλαίσιο των παγκόσμιων στοιχείων. 151 άνθρωποι στην Ευρώπη ε, πέθαναν λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων το 2014 παγκοσμίω. Ε, μιλούμε για πάνω από 32.000 θύματα. Να δούμε λίγο δηλαδή τη συνολική εικόνα θα έλεγα. Ε, γιατί θα ε, διαπιστώσουμε τότε ότι τα περισσότερα θύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Αυτό βεβαίως δεν αποτελεί λόγο να μην αναλάβουμε δράση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω διότι αναφερθήκατε και στη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Τι μάθατε, τι διδάγματα αντλήσατε από τα Panama Papers, διότι δεν αναδεικνύει το θέμα αυτό μόνο ότι πρόκειται για ε, φορολογικούς παραδείσους, για εκείνους που θέλουν να αποφύγουν την ε, φορολόγησή τους. Αντιθέτως, πρόκειται και για παραδείσους για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία γιατί είναι προφανές ότι το μικροέγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται με την τρομοκρατία. Και ποια είναι τα συμπαράσματα λοιπόν που αντλούν τα κράτη-μέλη από τις αποκαλύψεις των Panama Paper σε αυτό το θέμα. Επίσης, να σας ρωτήσω το εξής. Ανησυχώ με, σχετικά με τον όρο του, της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι όσον αφορά την συμμετοχή και την εμπλοκή συμπολιτών μας, των μουσουλμάνων στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος του τζιχαντιστή είναι προσβλητικός. Μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε για ψευδοθρησκευτικό, ψευδοθρησκευτική τρομοκρατία. Κάποιον άλλον όρο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευφύης η επιλογή ορολογίας που έχει γίνει. Ε, είναι κάπως ε, ε, αντιπαραγωγική η ορολογία που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τους ξένους μαχητές, τον όρο αυτών. Δική μας είναι. Δικό μας είναι το πρόβλημα. Είναι δικοί μας πολίτες, πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί που έχουν επιτεθεί στην Ευρώπη και σε άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε από αυτή την άποψη θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι επενδύσεις που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για την πρόληψη και την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης. Ιδίως αφού γνωρίζουμε, όπως είπατε κι εσείς, τη διασύνδεση με το μικρό και με το οργανωμένο έγκλημα και ότι οι φυλακές αποτελούν φυτόρια εκπαίδευσης τρομοκρατών. Τι γίνεται με, την, με τον κοινωνικό αποκλεισμό σε περιφέρειες των κρατών μελών μας. Κάτι που μπορεί να εξογήσει και την επιτυχία αυτών των εκστρατιών στρατολόγησης. Όσον αφορά την απειλή CBRN που επισημάνατε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της στρατηγικής CBRN γιατί το σχέδιο αυτό είχε ήδη αποδυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό από τα κράτη-μέλη εν συγκρίση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Κάποια κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν καθόλου, παρά μόνο τύπης. Και, όπως είπατε, υπάρχει και ένα συνδυασμός εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων πραγμάτων και φαίνεται για παράδειγμα ότι υπάρχουν διασυνδέσεις ακόμη και με οπλικά συστήματα τα οποία είχαν παραγγελθεί και από κράτη-μέλη και τη δική μου μεταξύ αυτών την Πορτογαλία. Φαίνεται ότι δεν είναι, δεν είναι πολύ σοβαρή η, η δράση που έχουν αναλάβει τα, κράτη, τα κράτη-μέλη. Τι γίνεται με τα βιολογικά ε, όπλα, πώς, τι θα γίνει με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που όλο και περισσότερα ε, διατίθενται και σε χαμηλές τιμές πλέον και τι γίνεται με τις απειλές όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Τέλος, για την κρυπτογράφηση. Είπατε ότι υπάρχει μια κατάχρηση της ανωνυμίας και της κρυπτογράφησης. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν μπορείτε να το ε, αποφύγετε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τραπεζικές συναλλαγές χωρίς κρυπτογράφηση, για παράδειγμα. Άρα, το ερώτημα είναι και το καθήκον είναι οι αστυνομικές αρχές να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικές και να προλαμβάνετε εσείς τους καλύτερους προκειμένου να αφοπλίζουν τους τρομοκράτες και προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς τα τεχνολογικά μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και τέλος, τι έχετε να πείτε για τους δίθεν συμμάχους μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που αποδεικνύεται ε, ε, ότι μάλλον άλλο ρόλο έπαιζαν. Μιλώ για την Τουρκία. Δημοσιογράφοι διώκονται διότι αποκαλύπτουν ότι η χώρα αυτή προμήθεσε το Ισλαμικό κράτος ε, με όπλα. Μιλώ για τη Σαουδική Αραβία. Για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται τον ε, ρόλο της χώρας αυτής και την βοήθεια που έχει δώσει σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Κυρία Ζήπα, ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Να ρωτήσω κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με τις διαφάνειες, που μας παρουσιάσατε. Έχουν συλληφθεί άτομα για τρομοκρατικές για εγκλήματα που συνδέονται με την τρομοκρατία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε συγκεκριμένα για τι είδους αδικήματα μιλούμε και τι είδους ε, αδικήματα έχουν διαπράξει αυτά τα άτομα. Είπατε επίσης για τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη διαφάνεια μας δώσατε αυτά τα στοιχεία. Πόσα δικαστήρια έχουν γίνει για αυτούς τους 513 ανθρώπους και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Οδήγησαν σε όλες τις περιπτώσεις οι διαδικασίες αυτές σε κυρώσεις, σε ποινές και ποια ήταν τα ακριβή αδικήματα για τα οποία επιβλήθηκαν ποινές. Επίσης, στις ε, εξηγήσεις που μας δώσατε, είπατε ότι γίνεται εκπαίδευση τρομοκρατών όχι μόνο στη Συρία, αλλά και σε βαλκανικές χώρες και ίσως, είπατε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. καλά, κατάλαβα. Υπάρχει δηλαδή εκπαίδευση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες και για συγκεκριμένους τόπους γεωγραφικούς όπου μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Για την αριστερή τρομοκρατία είπατε ότι είναι χαμηλού επίπεδου ε, έχετε αριθμούς και θα μπορούσατε να μας δώσετε και ορισμένε πληροφορίες σχετικά με το είδος των επιθέσεων που έχει κάνει η αριστερή τρομοκρατία. Για την ακροδεξιά τρομοκρατία μπερδεύτηκα λίγο. Είπατε ότι οι ακροδεξιές τρομοκρατικέ τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί. Είπατε ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των επιθέσεων, είπατε 9. Ταυτόχρονα όμως οι συλλήψεις που συνδέονται με ακροδεξιές τρομοκρατικές πράξεις έχουν μειωθεί. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την αντίφαση. Τώρα για τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είπατε ότι οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν ένα απόθεμα ε, εκρηκτικών μηχανισμών. Ε, καταλαβαίνω από αυτά που είπατε ότι προσπάθησαν χωρίς όμως επιτυχία. Ή είναι αλήθεια αυτό, καλά κατάλαβα ή έχετε πληροφορίες ότι ενδεχομένως να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Για την κρυπτογράφηση, πολύ σύντομα, γιατί το είπε και η Άννα εγώ κατανοώ ότι η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι η κατάχρηση της κρυπτογράφησης. Άρα η ίδια η κρυπτογράφηση δεν θεωρείται έγκλημα, ούτε θεωρείται στοιχείο ότι τη χρησιμοποιεί κανείς για να κρύψει κάτι και προσωπικά πρέπει να σας πω ε, ε, ότι έχω πιέσει για να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλο και περισσότερο την κρυπτογράφηση, όχι γιατί έχουμε κάτι να κρύψουμε, αλλά γιατί υπάρχουν πληροφορίες που είναι εμπιστευτικέ, Άρα χρειάζεται να χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση και ζητούμενο τώρα, τώρα είναι πώς θα καταπολεμήσουμε την κατάχρηση της ε, κρυπτογράφησης για την αποτροπή επιθέσεων. Αυτά. Ε, ο κύριος Σαρτζεντίνη. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους του Μόντους Operandi. Είπατε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ότι τα χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες, τις ροές προσφύγων οι τρομοκράτες για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει παρόλα αυτά κίνδυνος οι Σύριοι πρόσφυγες να ριζοσπαστικοποιούν ενώ είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ριζοσπαστικοποιηθούν ότι κυρίως από ντόπιο υλικό, είναι ντόπιοι οι τρομοκράτες που είχαμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο ρόλος των 200 ανθρώπων που προσλάβατε ή προσλαμβάνετε για να κάνετε τον έλεγχο στα hot spots. Πρόσληψη 200 ατόμων φαίνεται μεγάλος αριθμός, όμως έχουμε πολλούς που διέρχονται τα σύνορά μας. Άρα ίσως να είναι και λίγοι. Καταλαβαίνω θέλω να ξέρω κάποιες, ε, τι ακριβώς είναι τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι δουλειά κάνουν αυτοί οι 200 άνθρωποι. Όταν κάνουν αυτή τη διήθηση, αυτοί κάνουν τον έλεγχο των προσφύγων που καταφθάνουν. Στα κέντρα υποδοχής, στα hot spots, αλλού. Τι πληροφορίες συλλέγεται από αυτούς. Πώς σχετίζεται αυτό με τη δουλειά άλλων υπευθύνων, όπως των υπευθύνων για τους πρόσφυγες που εργάζονται στα hot spots. Ευχαριστώ, η κυρία Κιάνγκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατη. Ήθελα και εγώ ακριβείς πληροφορίες. Αν μπορείτε να τις δώσετε για ενδεχομένους κινδύνους για τους ανήλικους ε, που βρίσκονται όπου είναι το διαδίκτυο και που ε, ε, ριζοσπαστικοποιούνται μέσω του διαδικτύου και παιδιών, ανηλίκων τρομοκρατών. Μήπως υπάρχει κίνδυνος να προσιλητίζονται, να στατολογούνται ανήλικοι από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ κυρία Κέγκερ. Κυρία Ναβαρέτα, έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε αν έχετε την καλοσύνη Προσπαθήστε να απαντήσετε εντός ενός τετάρτου που έχει απομείνει για τη συζήτηση και προσπαθήστε να δώσετε απαντήσεις. Ορίστε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Yeah. Φαντάζεστε ότι από το 2016 που αυξάνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, το θέμα αυτό θα αποτελέσει επίκεντρο της συζήτηση και στην Ευρωπόλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όπως σας είπα, εμείς συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, τις ε, ε, συμπιλίζουμε, συγκεντρώνουμε πληροφορίες και από τους οργανισμούς στο ΤΕΣΑΤ και προσπαθούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και να διαμορφώσουμε μία εικόνα. Αυτό έγινε για το 2015 για να αξιολογήσουμε την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, οι περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις, περίπου το 90% αυτών, ε, είναι τζιχαντιστικές, τζιχαντιστικής τρομοκρατίας. Μάλιστα, σε συζητήσεις που κάναμε τα κράτη-μέλη, ε, καταλάβαμε ότι η έννοια της διχατιστικής τρομοκρατίας μπορούν να, στην αρχή να ήταν κάπως αόριστη και αφήσιμη. Γιατί ακριβώς αυτοί οι τρομοκράτες ε, χειραγωγούν το Ισλάμ και έναν από τους ε, πυλώνες του Ισλάμ που είναι ο Ιερός Αγώνας, Τζιχάντ. Και έτσι προσπαθούν να προωθήσουν την εξτρεμιστική τους αυτή θεώρηση της θρησκείας της Ισλαμικής. Και προσπαθούν να κηρύξουν αυτόν τον ιερό αγώνα ή καπηλεύονται τον ιερό αγώνα για... και το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την τρομοκρατία, για την προσπάθειά τους, την τρομοκρατική. Και μάλιστα στην προσπάθεια αυτή ορισμού της τρομοκρατίας ε, συμμετέχει και η Europol στη συζήτηση. Και προσπαθήσαμε να έχουμε μια πιο ε, συμπαγή προσέγγιση σε αυτή τη διχατιστική τρομοκρατία. Και Γι' αυτό και έχουμε σε αυτή τη μονάδα μας ε, ανοιχτή συζήτηση με τα κράτη-μέλη για να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το θέμα και να βρούμε έναν τρόπο όταν μιλούμε για την τρομοκρατία να ξέρουμε τι εννοούμε. Τώρα το ότι χρησιμοποιούμε και το τζιχαντιστικό ω επίθετο δεν έχει σημασία γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομοκράτες πραγματικά. Τώρα πώς εξελίσσεται αυτή η τρομοκρατική απειλή. Ε, είναι πρωτοφανής ε, αυτή η ραγδαία εξέλιξη. Γιατί από την τρομοκρατία πολλά κρατημέλη υπέφεραν εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι το 2015 είχαμε όμως κάποιες επιθέσεις, αλλά με μονομένων ε, φορέων των μοναχικών καβαλάριων. Βέβαια, όσο γενικεύεται η εκπαίδευση, τόσο πιο θανατηφόρο είναι το πλήγμα της τρομοκρατίας. Γιατί γίνεται πιο οργανωμένη. Και σε αυτές τις εμπόλεμες ζώνες στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ παρέχεται εκπαίδευση και ε, υπάρχουν και ικανότητες και πόροι για να γίνουν πιο θανατηφόρες, πιο επικίνδυνες αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις και πιο προσαρμοσμένες στο τοπικό περιβάλλον. Ήταν ραγδαίες λοιπόν αυτές οι εξέλιξεις και είδαμε αυτές τις προσαρμογές ε, στη Γαλλία και στο, στο Παρίσι δηλαδή και στο Βέλγιο. Και είδαμε πως ε, τρομοκράτες από τη Συρία, από το Ιράκ είχαν διασυνδέσεις με τρομοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί μάλιστα είχαν ε, εμπειρία από την εκπαίδευσή τους στην Συρία και το Ιράκ. Και αυτός ο συνδυασμός και αυτή η συνεργασία τους κάνει ακόμη πιο αποτελεσματικούς και θανατηφόρους στις ενέργειές τους. Και το είδαμε αυτό το 2015. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσης, φαίνεται ότι διευκολύνει την εξάπλωση της τρομοκρατίας. Γιατί έτσι μπορούν να εντοπίσουν τους ευάλωτους στόχους τους. Επίσης, ε, έτσι ε, διαδίδουν καλύτερα και πιο εύκολα το το μήνυμά τους. Γι' αυτό και η, ριζοσπασ... η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης είναι πιο σύντομη πια, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, βλέπουμε ότι εστιάζονται σε συγκεκριμένους στόχους, πιο ευάλωτους γυναίκες, αναφέρθηκε κιόλα, γιατί πιστεύουν ότι και οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν ε, ιδιαίτερο ρόλο στις ομάδες αυτού του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Και Γι' αυτό προσπαθούν να στρατολογήσουν και οι γυναίκες στη Συρία και το Ιράκ. Επίσης έχουν αναπτύξει ειδική προπαγάνδα για τους νέου. για να έχουν περισσότερη απήχηση στους νέου. Έχουμε ακόμη και ανήλικες, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν περισσότερο, οι νέοι, ε, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοια προπαγανδιστικά μηνύματα και θα πρέπει να βρούμε μέτρα για να αποτρέψουμε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση. Να δώσουμε ένα εναλλακτικό, σε ένα, ε, εναλλακτική ρητορική και να μειώσουμε την έκθεσή τους σε αυτά τα απλά αλλά ισχυρά μηνύματα. Και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Η Αλκάιδα δεν χρησιμοποίησε πολύ τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κυρίω ε, να προωθήσει τη βία, να την εξυμνήσει, να τη δικαιολογήσει και να εξυμνήσει τους οπαδούς τους. Το Ισλαμικό μα κράτο είναι πιο πρακτικό, γιατί εξακολουθούν να στέλνουν ένα όχι μόνο θρησκευτικό μήνυμα, είναι βέβαια ακόμη θρησκεία στο μήνυμα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά θρησκευτικό το μήνυμα. Έχουν διευρύνει το μήνυμά τους και είναι πιο ανοιχτοί. Προσπαθούν να προσελκύσουν και άλλους προκειμένου να βοηθήσουν το Ισλαμικό κράτος. Δεν περιορίζεται λοιπόν μόνο στο θρησκευτικό χαρακτήρα του μήνυματος. Και στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού και των Βρυξελών το είδαμε. Δεν είναι πια οι μοναχικοί καβαλάριδες αυτοί που κάνουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουμε πιο οργανωμένο φαινόμενο τρομοκρατίας. Επίσης, Είχαμε κάποιον που με ένα μαχαίρι πήγε και μαχαίρωσε τρεις στρατιωτικούς ε, στην Ίκαια. Μετά από κάποιες προπαγανδιστικές πληροφορίες που άκουσε για το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολύ, πολλές μορφές ε, αυτής της, της βίας που συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος. Επαναλαμβάνω, έχουν στο στόχο αυτό τους και ειδικές κατηγορίες γυναίκες, νέους. Χρησιμοποιούν μάλιστα στην προπαγάνδα τους όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν έχουν μόνο προπαγάνδα στα αραβικά. Έχουν α, πληροφορίες και στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, απευθυνόμενοι σε πολύ ευρύτερο κοινό πια. Και στις προσπάθειες που κάνουμε είναι να προωθήσουμε και στο διαδικτύο κάποιες δραστηριότητες πανευρωπαϊκά. Τώρα γιατί λέω να προωθήσουμε περισσότερο σε Ευρωπαϊκή Ένωση παρά ως κρατη Θα πρέπει να συνδυάσουμε και να συσπηρώσουμε τις προσπάθειές μας με τα κρατη και με την Ευρωπόλ για να καταπολεμήσουμε και διαδικτυακά την τρομοκρατία. Και μάλιστα με τη μονάδα αναφορά ψηφιακού περιεχομένου έχουμε και εθνικέ ομάδε και εθνικά σημεία επαφή για να καταπολεμήσουμε την διαδικτυακή προπαγάνδα των τρομοκρατικών ομάδων. Και τα περισσότερα κρατημέλη έχουν αντίστοιχε ομάδε αναφορά ψηφιακού περιεχομένου, αντίστοιχη με την IRU που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε επαφέ με εμπειρογνώμονε. Και μάλιστα δεν γίνεται απλώ έλεγχο του διαδικτύου, γιατί έχουμε αυτή την πρωτοβουλία από το 2008 του Check the Web, μια γερμανική πρωτοβουλία για να γίνει μια αφύπνιση της τρομοκρατικής ε, αξιοποίηση του διαδικτύου. Τέτοιες πρωτοβουλίες πια υπάρχουν σε πολύ περισσότερα κράτη. Το βασικό όμως είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη, γιατί η Ευρωπόλη είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μόνο. Και έχουμε τους καλύτερους εμπειρογνώμονες ε, στη Χάγη και προσπαθούμε να συστήσουμε μια διατομεακή προσέγγιση με εμπειρογνώμονες ώστε να εμπλουτίσουμε την εργαλειοθήκη μας για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την τρομοκρατία, συμπεριλαμβάνοντας και την πρόληψη στα εργαλεία μας και φυσικά θέλουμε καλύτερη διασύνδεση με τα κράτη-μέλη. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια νέα φωνή και καλύτερη συνεργασία για να γνωρίζουν τα κράτη-μέλη πώς χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο. Μόνο γνωρίζουμε τα μέσα τους μπορούμε να τα κατατροπώσουμε και να δούμε να προστατεύσουμε τους πιο, τις πιο ευάλωτες ομάδες. Θέλουμε νέα φωνή και στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση και ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη διαδικτυακή τρομοκρατία. Όσον αφορά την διασύνδεση παράνομης μετανάστευσης και τρομοκρατίας. Οι τρομοκράτες είναι τυχοδιώκτες. Χρησιμοποιούν κάθε μέσο, οτιδήποτε έχουν στη διάθεσή τους για να προωθήσουν τους δικούς τους στόχους. Και η χρήση, η αξιοποίηση δηλαδή αυτών των ροών ανθρώπων που έρχονται μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη από τη Συρία και, και το Ιράκ είναι ε, μια ευκαιρία που θα την αξιοποιήσουν κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχουμε βρει ακόμα συστηματικά στοιχεία ε, ε, ότι το κάνουν, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι έχει συμβεί αυτό. Και Κάποιοι από τους ανθρώπους που ε, ε, εμπλέκονται και στις επιθέσεις του Παρισιού ε, σχετίζονται και με αυτές τις προσφυγικές ροές. Και υποστηρίζουμε και την Ιταλία και την Ελλάδα σε σχετικές δραστηριότητες που έχουν αναλάβει για τον αντοπισμό τέτοιων ατόμων. Σκοπός της Europol είναι να, να δώσει υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Εμείς εργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες και συνεργαζόμαστε, παρέχουμε βοήθεια στους Ιταλούς και Έλληνες συναδέλφους μας, ακριβώς για να αντιμετωπιστεί η απειλή. Όσο περισσότερο καταπολεμούμε την εγκληματικότητα και την ε, εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ανθρώπων προς την Ευρώπη, τόσο αποτελεσματικότεροι θα γίνουμε και όσον αφορά την ε, αποτροπή της τρομοκρατικής απειλής. Είναι συνδυασμός πραγμάτων δηλαδή. Η ασφάλεια συνδέεται και με την καταπολέμηση των δρομοκρατικών ε, δικτύων και της αξιοποίησης, της εκμετάλλευσης των ε, θυμάτων, των διπλών θυμάτων, των προσφύγων δηλαδή, ακριβώς διότι χρειάζεται αφενός, είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και σε δεύτερη φάση γίνονται θύματα των ε, τρομοκρατικών δικτύων. Ξαναλέω, δεν έχουμε συστηματικές ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο γίνεται, αλλά γνωρίζουμε ότι σε έναν βαθμό συμβαίνει και αυτό και στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας στα hot spot, στα νησιά στην Ελλάδα και στη Σικελία, στην Ιταλία, σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Frontex και κινητήρια δύναμη σε αυτές τις δραστηριότητες είναι πάντοτε τα κράτη-μέλη. Εκείνα είναι αυτά που αποφασίζουν για το τι δράσεις πρέπει να αναλυφθούν όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια άτομα που έρχονται μέσω αυτών των προσφυγικών ροών στο έδαφος τους συνδέονται με την τρομοκρατία. Και δύο ακόμη στοιχεία που θέλω να πω αφορά, ε, αφορούν την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πώς συμβαίνει, πώς γίνεται αυτή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο ρόλος της αδελφότητας στη Γαλλία και στο Βέλγιο ε, ήταν ένα, μια αφορμή για να δώσουμε στοιχεία ή για να ε, εξάγουμε κάποια στοιχεία ε, για το τι συμβαίνουν, συμβαίνει ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Συνήθως όμως τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι αυτοί ε, μετρητά. Βρισκόμαστε ακόμη σε συζητήσεις με τους Γάλλους και βέλου συναδέλφους μας για να, δια... να εξακριβώσουμε πώς ακριβώς χρηματοδοτήθηκαν αυτές οι επιθέσεις, ποιος τις συνέλαβε, ποιο τις χρηματοδότησε και ποιος κατήφθηνε την ε, αξιοποίηση των χρημάτων για τη διάπραξη αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Έχουμε ακόμα στοιχεία ε, που μας λείπουν, αλλά γι' αυτό ε, άλλωστε συνεχίζουμε τις έρευνες για την ακροδεξιά τρομοκρατία. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Ελπίζω στο, στην ιστοσελίδα μας να δημοσιευθούν αυτά σε δύο-τρεις εβδομάδες. Όσον αφορά τώρα την ακροδεξιά τρομοκρατία όμως, Οι επιθέσεις έγιναν το 2015 κυρίως στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Αναφέρονται 9 επιθέσεις. Δεν υπήρξαν θύματα. αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για αύξηση σε σύγκριση με το 2014. Και αυτό δεν συνδέεται με τις συλλήψεις. 33, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια αντιστοιχία με τις ε, συλλήψεις. Από 33, 11. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι πολλές από τις έρευνες ε, ε, έγιναν πριν από το 2014 και οι συλλήψεις έγιναν το 2014 αλλά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ μεγάλο βάθος λεπτομέρειας για να εξετάσουμε από πού προήλθε αυτό, αυτός ο αριθμός το 11 το 2015. Στην, το 2015 ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση ακροδεξιάς τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Οι περισσότερες ε, επιθέσεις έγιναν στην Ισπανία, 4, Ιταλία 3 και Ελλάδα 2 αυτός είναι μεγαλύτερος αριθμός από ό,τι καταγράφηκε το 2014, αλλά όπως είπα, στην ιστοσελίδα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιευτούν όλα αυτά τα στοιχεία αναλυτικότατα. Και κάτι τελευταίο που αφορά τον καταδικαστε, τους, τους καταδικαστέντες. Εγώ δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή μαζί μου για να σας πω πόσοι καταδικάστηκαν. Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν στην TSAT αυτά τα στοιχεία Α, συγγνώμη, κάτι έχω τελικά. Το 2015, 12 κράτη-μέλη ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρώσει 208 δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Αλλά θα έπρεπε να το αναλύσω αυτό το στοιχείο για να σας πω πόσοι τελικά καταδικάστηκαν και πόσοι αθώθηκαν αλλά όπως είπα, πολύ σύντομα θα έχετε στη διάθεσή σας τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ναβαρέτε. Να σας ευχαριστήσω για τις αναλυτικές απαντήσεις που μας δώσατε. Ε, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες και σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Πρέπει να περάσω αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερής σας διάταξης. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, τελευταίο σημείο για σήμερα, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου και την Κομισιόν. Η Κομισιόν παρουσίασε στις 4 Μαΐου ε, με βάση το άρθρο 29 μια πρόταση ε, για σύσταση ε, προσωρινού ε, ελέγχου εσωτερικών συνόρων σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτει σε κίνδυνο την ε, συνολική λειτουργία του, ε, της, του χώρου Σέγγεν. Η σύσταση αυτή υιοθετήθηκε στις 12 Μαΐου και από την ημερομηνία αυτή η Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία μπορούν να συστήσουν ε, προσωρινούς συνορικούς ελέγχους για ανώτατο διάστημα έξι μηνών σε συγκεκριμένα σημεία των εσωτερικών συνόρων. Θα, ακούσουμε την ε, Προεδρία του Συμβουλίου και στη συνέχεια την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ο κύριος Λούστερμπουργκ έχει το λόγο εκ μέρους της Ολλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής που μας δίνουν ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη σύσταση του Συμβουλίου αναλυτικά. Πράγματι είναι εφαρμοστική απόφαση που θέτει το Συμβούλιο στις 12 Μαΐου και καθορίζει μια σύσταση για προσωρινούς εσωτερικούς μεθορικούς εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Αυτή η σύσταση του Συμβουλίου είναι συνέπεια αυξανόμενου αριθμού μεταναστών που εισήρχονται στην περιοχή Σέγγεν, κάτι που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι και αυτό οδήγησε σε αποφάσεις αρκετών κρατών μελών προσωρινά να επανισάγουν εσωτερικούς μεθοριακούς ελέγχους σε κάποια τμήματα των εσωτερικών συνόρων για λόγους δημόσιας πολιτικής. Αυτοί οι εσωτερικοί μεθορικοί ελέγχοι εισήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες του κεκτημένου Σέγγεν και ήταν περιορισμένοι οι έλεγχοι χωρικά και χρονικά. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Επιστροφή στο Σέγγεν» του η Μαρτίου ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα που υπάρχει μιας προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των προσωρινών μαθηριακών ελέγχων μετά μια περίοδο της 12 η Μαΐου, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο και πράγματι στις 4 Μαΐου παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση βάσει προσεκτικής αντελεχούς αναλύσεως που συνεπέρανε ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρές ελλείψεις σε κάποια τμήματα των εξωτερικών συνόρων Σέγγεν που θέλουν σε κίνδυνο τη γενική λειτουργία της περιοχής Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν. Αυτή η πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου έχει στόχο τη συνέχιση εσωτερικών μεθοδικών ελέγχων από τα πέντε κράτη-μέλη που αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, που διενεργούν εσωτερικού ε, μεθοριακού ελέγχου για του λόγου, επαναλαμβάνω. Αυτό αφορά την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Νορβηγία. Το Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ότι θα πρέπει να ενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι σε αυτά τα τμήματα εσωτερικών συνόρων που θεωρείται ότι αυτό είναι αναγκαίο και είναι αναλογικό μέτρο. στι 12 Μαου. το Συμβούλιο υιοθέτησε αυτή την εφαρμοστική απόφαση και δημιουργείται εξ αυτού η σύσταση ενώ μεταξύ μετά την υιοθέτηση και η Γερμανία και η Αυστρία κοινοποίησαν προς το Συμβούλιο ότι απεφάσισαν να συνεχίσουν τους εσωτερικούς τους μεθοριακούς ελέγχους βάσει της συστάσεως. Αυτά από την πλευρά μου και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λίστερμπορκ. Η κυρία Μος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά από τη δική μας κοπιά, γιατί εκπρόσωπος του Συμβουλίου εξήγησε λεπτομεριακά τα διάφορα βήματα. Ίσως ένα συμπληρωματικό στοιχείο, όπως αναφέρεται στο δικό χάρτη επιστροφή στο Σέγγεν, στόχος μας είναι να επανέλθουμε στο χώρο του Σέγγεν χωρίς εσωτερικούς ελέγχους των συνόρων προς τα τέλη του έτους, του τρέχοντος έτους. Μάλιστα αναγνωρίζουμε τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια, η Ελλάδα επικουρήθηκε και από τεχνική και οικονομική συνδρομή και από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τα κράτη-μέλη και έχει σημειώσει πρόοδο σε θέματα ε, διαχείριση του ελέγχου των συνόρων. Επίσης, ε, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ήδη έχει αποφέρει τους πρώτους καρπούς. Βέβαια, το Συμβούλιο συμφώνησε και είναι υπέρ της σύστασης. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά σύνορα στα οποία τα δίνονται να εφαρμόσουν ακόμη ελέγχους, θα πρέπει να γίνονται με τρόπο αναλογικό και όσο είναι απολύτω απαραίτητη αυτή η έλεγχη στα εσωτερικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και θα έχει και τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για να μπορεί να διαπιστώνει πώς έχουν τα πράγματα επί τόπου. Ευχαριστούμε κυρία Μασχάμερ. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ. Uh, Όχι, άρα ήταν όλα φως φανάρι, μας τα εξηγήσατε πολύ καθαρά και με σαφήνεια. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε στην Επιτροπή μας και μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο από τις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη συνεργασία σας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για τη διερμηνία τους. Ραντεβού αύριο στις 9. Καλό σας απόγευμα.